τους συναδέλφους. Χαίρομαι που μας ακούτε όσοι μας ακούτε. Το θέμα μας είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων. Έχουμε προσκαλέσει ορισμένα άτομα ειδικά. Υποθέτω ότι η συζήτηση θα πολύ ενδιαφέρουσα. Με διάφορες παρουσιάσεις. Έχουμε και εκπρόσωπο της Επιτροπής. Έχουμε το δίκτυο Impel με τον ε, Jack McLean που είναι διευθυντής Jacqueline McLean Τη Jacqueline λοιπόν έχουμε ένα σύνολο μιλητών υψηλού επίπεδου Θέλω να δώσω το λόγο καταρχήν στον εκπρόσωπο της Επιτροπής εν συνεχεία στους υπόλοιπους ε, ομιλητές του πάνελ και στο τέλος στους ε, συναδέλφους που είναι παρόντες. Βλέπω εδώ πέρα ότι οι σοσιαλιστές είναι υπερεκπροσωπούνται. Θα μπορούσαμε σχεδόν να κάνουμε συνεδρίαση ομάδας. Τι ωραία. Είναι μόνο σοσιαλιστές εδώ πέρα. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ, κύριε μου στον κύριο. Χούλιο Αθίαμπορτες, Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Κομισιόν να παρουσιάσει σήμερα την έκθεσή της για την εφαρμογή του καονισμού για την αποστολή των αποβλήτων. Στην παρουσίασή μου να εξηγήσω καταρχήν τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Με συνεχεία να διευκρινίσω το πεδίο, την εμβέλεια της έκθεσης και συνεχεία να σταθώ σε κάποια από τα βασικά πορίσματά της. Καταρχάς, η μεθοδολογία. Τρίτη έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή της, του κανονισμού για την αποστολή αποβλήτων ε, δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 51 του κανονισμού και καλύπτει τα έτη 2007, 2008, 2009. Η έκθεση βασίζεται σε δύο διαφορετικές εκθέσεις που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη-μέλη σε αιτήσια βάση. Η πρώτη είναι ένα αντίγραφο της έκθεσης στην γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας που έχει ποσοτικά στοιχεία για τις διασυνοριακές κινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων. Η δεύτερη έκθεση προβλέπει να σταλούν περαιτέρω πληροφορίες προς την Κομισιόν, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια. Οι υποβολές των εγγράφων των κρατών γίνεται ηλεκτρονικά στη Eurostat. Εν συνεχεία η Eurostat ετοιμάζει πίνακες και αριθμητικά στοιχεία που μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο το εσωτερικό της Κομισιόν που δημοσιεύεται, μαζί με την έκθεση και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος συντάσσει το κυρίως κείμενο της έκθεσης. Η γενική στατιστική εικόνα που προκύπτει από την έκθεση είναι αξιόπιστη κατά την άποψή μας. Ξέρουμε βεβαίως ότι υπάρχουν κάποια κενά και διαφορές, ανακρίβειες που οφείλονται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, η καθυστερημένη υποβολή των εκθέσεων από κάποια κράτη-μέλη. Δεν θα τα κατανομάσω, τα κρατη που καθυστέρησαν. Αναφέρονται όμως το κείμενο της έκθεσης. Είναι προφανές ότι αν τα κράτη-μέλη δεν αναφέρουν τα δεδομένα που πρέπει να αναφέρουν, η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης. Σε ορισμένε περιπτώσεις, η Eurostat μπόρεσε να κάνει εκτιμήσεις για να καλύψει κάποια κενά. Δεύτερον, Υπάρχουν κάποιες ε, προφανείς διαφορές στα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη, διαφορές και ανακρίβειες. Λογικά το συνολικό νούμερο για τις εισαγωγές και εξαγωγές ε, αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Με βάση τα δεδομένα που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη, οι εξαγωγές εκτός ενός κρατούς μέλους είναι υψηλότερε από τις εισαγωγές. Για το πεδίο εφαρμογή. η έκθεση της Κομισιόν παρουσιάζει δεδομένα σε ό,τι αφορά την δημιουργία ε, σκουπιδιών και την διασυνοριακή κυκλοφορία ή μετακίνηση επικίνδυνων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν καλύπτει ε, την ε, διασυνοριακή κίνηση μη επικίνδυνων ουσιών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης ή κοινοποίησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση με βάση την κοινοτική νομοθεσία να αναφέρουν τα κράτη-μέλη αυτές τις κινήσεις. Συνειδητοποιούμε όμως ότι είναι σημαντικό να έχουμε εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των αποστολών αποβλήτων ακόμα και όταν τα απόλυτα αυτά δεν είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την, πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που παρακολουθεί ε, τις κινήσεις αποβλήτων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και εκτός, γιατί κάνει μια πλήρη ανάλυση ε, μη επικοινωνουσιών, δεδομένα, εξαγωγές μετάλλων, χαρτιού και πλαστικών αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Για τα πορίσματα της έκθεσης υπάρχουν τέσσερις πτυχές που θα ήθελα να τονίσω. Καταρχήν, η αύξηση στα επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούν που προέκυψαν ανάμεσα στο 2000 και στο 2008 τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 46%. Το 2009 είχαμε μία μικρή μείωση, αλλά αυτό μάλλον οφειλόταν στην οικονομική κρίση. Η αύξηση σε επικίνδυνα απόβλητα δείχνει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων για την επεξεργασία. Ε, είναι σημαντικός ο ρόλος της τρίτης χώρας. Το 2009 πάνω από 50% 90% όλων των επικίνδυνων ουσιών ε, έτυχαν επεξεργασίας στη χώρα όπου δημιουργούνται τα απόβλητα. Χώρες όμως όπως το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία έχουν υψηλά ποσοστά εξαγωγής πάνω από το 40%. Μερικές από αυτές τις χώρες, η Ολλανδία ας πούμε και το Βέλγιο, εισάγουν σημαντικά ποσά επικίνδυνων ουσιών. Τρίτο πόρισμα. Από όλα τα πιο... Από όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που τα επεξεργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αύξηση των διασυνοριακών κινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ειδικά από το 2001 και μετά. Έχουμε την αρχή της γειτονίας εδώ, την ε, λαμβάνουμε υπόψη μας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη όμως υπάρχουν ε, πολύ προηγμένες ε, εγκαταστάσεις για την επεξεργασία επικίνδυνων ουσιών που λείπουν σε άλλα κράτη-μέλη. Και συχνά για πολλά κράτη-μέλη οι πιο η πλησιέστερη εγκατάσταση βρίσκεται σε ένα άλλο κρατό μέλο, Δεν υπάρχει καν στο δικό τους. Κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον ακόμα. Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά επιτύχει την αυτάρκεια στην επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή να βασιστούμε στο δυναμικό που έχουν τρίτες χώρες. Πάνω από το 90% όλων των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων ουσιών ε, λαμβάνουν χώρα μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό τέτοιων ουσιών, τέτοιων αποβλήτων αποστέλλεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει καθαρός εισαγωγέας επικίνδυνων ουσιών και από το 2001 οι εισαγωγές ήταν 5 με 10 φορές υψηλότερες από τις εξαγωγές. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι οι εμπορικές ροές για τις επικίνδυνες και μη επικίνδυνες ουσίες και απόβλητα πηγαίνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρός εξαγωγέας μη επικίνδυνων αποβλήτων και καθαρός εισαγωγέας επικίνδυνων αποβλήτων. Πάμε τώρα στις παράνομες μεταφορές αποβλήτων ή αποστολές αποβλήτων. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα, ένα μεγάλο... ένας άγνωστος χ. Η νομοθεσία μας απαγορεύει κάποιες αποστολές επικίνδυνων ουσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και αποβλήτων προς διάλυση σε χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΖΕΣ, αυτές οι αποστολές απαγορεύονται. Αν κοιτάξουμε τα επίσημα νούμερα, εύκολα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι παράνομες αποστολές δεν παίζουν σημαντικό ρόλο Μόνο 400 περιπτώσεις παράνομων αποστολών αναφέρθηκαν για το 2009. Ξέρουμε όμως ότι, ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου και οι επιθεωρήσεις που κάνει η Ιμπελ δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές παράνομες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τις επιθεωρήσεις αποστολών αποβλήτων. Πιστεύουμε... Αυτό αναφέρεται στην εκθεσή μας. Αξιολογούμε τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και θα υποβάλουμε του χρόνου μια νομοθετική πρόταση για να ενισχύσει τις προϋποθέσεις ε, επιθεωρήσεων στον κανονισμό για τις αποστολές αποβλήτων. Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις ροές επικίνδυνων αποβλήτων που συνδέονται με τις παράνομες εξαγωγές, ας πούμε. Παραδείγματο χάρη ε, οχήματα στο τέλος της ζωής τους και ηλεκτρονικά αποβλήματα, απόβλητα. Για τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουμε μια νέα οδηγία που έχει αποδείξει το βάρος απόδειξης. Ε, βαραίνει τον εξαγωγέα αυτό το βάρος, δηλαδή ο εξαγωγέας χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού υλικού θα πρέπει να δώσει απόδειξη, αποδεικτικά στοιχεία ότι τα υλικά αυτά δεν είναι ηλεκτρονικά. Για, για την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος ζωής τους, οι κατευθυντήρες γραμμές για την αποστολή αποβλήτων, δηλαδή οχημάτων που είναι απόβλητα, έχουν ε, δημιουργηθεί μαζί με, τους, ε, με τις χώρες που εξάγουν τέτοια απόβλητα. Και αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές εφαρμόζουμε ήδη, ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011. Όλα όσα είχα να πω ήταν αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω τα πορίσματα της έκθεσης να είναι χρήσιμα για τη δουλειά που κάνουμε πάνω στα απόβλητα και τις κινήσεις αποβλήτων. Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε και θα ακούσω όποιες υποδείξεις έχετε να μου κάνετε για να βελτιώσω το μηχανισμό ε, υποβολής εκθέσεων. Ο πρόεδρος κ. Γκρότε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του θέματος. Η έκθεση τώρα της διευθύντριας της EA Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Θα πρέπει να βρήκατε αντίγραφο της έκθεσης που έχουμε ετοιμάσει για διαχείριση και τα μετακίνησει αποβλητών στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σας έκανε μια παρουσίαση για να σας πει ε, τι έχει γίνει σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο και να δούμε ποιε είναι οι τάσεις που δημιουργούνται εδώ πέρα. Να ε, δούμε τι γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Υπάρχουν ενδιαφέροντες αριθμοί. Εάν σκεφτείτε τι έγινε στα τελευταία 10 και 20 χρόνια, ε, από το 1990 ως το 2011, οι εξαγωγές αποβλήτων λόγω χάρη για το ε, αλουμίνιο, το νικέλιο, το χάλιβα και το σίδηρο έχει αυξηθεί. Τα απόβλητα από μέταλλα και πλαστικό έχουν πενταπλασιαστεί. Αυτή είναι σημαντική αριθμή εάν σκεφτεί κανείς ε, την εμβληματική πρωτοβουλία που θέλουμε για την ε, διαχείριση των ε, αποβλήτων. Επίσης, ο όγκο των αποβλήτων διπλασιάστηκε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία για όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε πρέπει να δούμε γιατί αυξάνονται τα απόβλητα και πού κατευθύνονται. Ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρει για την διασυνορική ε, μετακίνηση των αποβλήτων είναι το κατά πόσον αυτά οδηγούνται σε ε, ε, διάθεση ή σε ανακύκλωση στις χώρες όπου καταλήγουν. Είναι θετικό το στοιχείο αυτό αν υπάρχουν προβλέψεις γι' αυτό με, από την άποψη του περιβαλλοντικού και του οικονομικού κόστους. Επίσης τα απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν ως πόρος για την παραγωγή. αυτό είναι καλό εφόσον δεν ανατρέχουμε σε πρώτε ύλε που δεν έχουν ξανά Είναι πολύ σημαντικό από την άποψη τη πολιτισματική διαχείριση των πόρων για την οικονομία. Όμω υπάρχουν κίνδυνοι ω προ τι μεταφορέ, τι περιβαλλοντικέ ε, δυσκολίε και βεβαίω πλέον σημαντικό η χώρα προορισμό. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε με βάση την έκθεση αυτή και μέσω των ε, όσων κάνει η Ερμοδία Επιτροπή, είναι να δούμε κατά πόσον μπορούν αυτοί που τα παραλαμβάνουν να τα διαχειριστούν και μάλιστα με ασφάλεια. Αυτό που μας απασχολεί λοιπόν είναι ακριβώ τι γίνεται με τα προϊόντα που καταλήγουν σε μια χώρα όπου δεν υπάρχουν καθόλου εγκαταστάσει ή ακατάλληλε εγκαταστάσει. Θα το ξαναδούμε αυτό. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση την περίοδο που καλύπτει η συγκεκριμένη έκθεση. Η δημιουργία και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς από το 1993 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει και την διασυνοριακή ε, μετακίνηση όλων των αγαθών συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων. Όμως οι ε, πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει μεριδώσει και εναλλακτικά προϊόντα. Υπάρχουν λοιπόν καλοί, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα απόβλητα στον όγκο του Ταυτόχρονα έχουμε και πολλούς εναρμονισμένους και κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτοί απλώ απαιτούν νέε προσεγγίσει για την διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων. Έχουμε αποφύγει την διάθεση των αποβλήτων στι κομματερέ και έχουν καταλήξει σε διαδικασίε ανακύκλωση τα απόβλητα αυτά. Κάποιε φορέ οι εγκαταστάσει επίση πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου υπ' αυτή τη σκοπιά. Γι' αυτό λοιπόν ε, όπου δεν υπάρχουν εγκαταστάσει ε, υπάρχουν εξαγωγέ αποβλήτων από τη μια χώρα σε άλλη. Και αυτό μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση. Υπάρχουν επίση και μη ρυθμιστικοί παράγοντε που συντελούν εδώ, όπω η οικονομική ανάπτυξη σε κάποιε χώρε, ε, που ζητούν περισσότερε ύλε. Η Ασία είναι κατεξοχήν ε, προορισμό για πλαστικέ ύλε. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Επίση, για την παραγωγή ενέργεια. Επίση, πολλά πράγματα καταλήγουν σε αποτευρωτήρε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποιες είναι, ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα εδώ. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με τις κατηγορίες των αποβλήτων. Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ των διαφόρων ειδών αποβλήτων. Οι επικίνδυνες ουσίες λόγω χάρη, που είναι ένα μεγάλο ε, ποσοστό των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Υπάρχουν όμως διαφορές μεταξύ της ε, εθνικής, της εθνικής δυνατότητας κάθε να τα διαχειριστεί αυτό καθορίζει και τι συνορικέ μετακινήσει των αποβλήτων. Υπάρχουν ε, διαφορέ στο κόστο ανάκτηση, διαφορετικοί προορισμοί. Κάποιε φορέ ο προορισμό είναι εντό των σύνορων, κάποιε λίγο πιο μακριά από τα σύνορα. Είναι λοιπόν σημαντικό και παράγοντα του κόστου. Επίση για τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν σοβαρές ποσότητες που κατευθύνονται εκτός ε, Ευρώπης, όπως τα πλαστικά που ανέφερα στην Ασία και άλλες ε, κατηγορίες. Αυτό είναι μια ένδειξη για το που υπάρχει ζήτηση για συγκεκριμένους πόρες και ε, που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν. Και πέραν από τους στόχους της ανακύκλωσης, τι μας δείχνουν όλα αυτά, ότι Πραγματικά οι στόχοι της ανακύκλωσης με τις οδηγίες ε, για τα απόβλητα έχουν δώσει μεγαλύτερα κίνητρα. Δημιουργείται μια νέα αγορά με νέα προϊόντα. Η διάθεση ανανεώσιμων, ανακυκλώσιμων μάλλον ε, πόρων πλέον είναι ένα στοιχείο που εδώ συμβάλλει στην συνολική εικόνα. Για την ε, εξαγωγή λόγου χάρη, χάλιβα και παλιοσίδερου. Είδαμε μια μεγάλη αύξηση το 2011. Βλέπουμε ένα σημαντικό 8 δις ε, συνολικά όγκο. Πρέπει να δούμε τώρα τι, οικονομική, οικονομικό κέρδος εδώ έχουμε και αν υπάρχει και ζημιά για το περιβάλλον. Θα ήθελα να μιλήσω και για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία συνήθως θεωρούνται επικίνδυνα, είναι παράνομα, εάν αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες εκτός ΩΣΑ. Και το θέμα είναι πώ καταγράφονται στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εκεί φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατευθύνονται προ την Δυτική Αφρική, την Ασία, αλλά με την ετικέτα των μεταχειρισμένων αγαθών. Αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα εδώ. Ένα μεταχειρισμένο προϊόν θα μπορούσε ενδεχομένω να διορθωθεί, να επισκευαστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί στην Ασία. Έχει ένα κύκλο ζωή όμω και σε αυτή τη χώρα και θα καταλήξει έναν απόβλητο. Δηλαδή το πρόβλημα δεν αποφεύγεται, ούτε επιλύεται, απλώ αναβάλλεται η επίλυσή του. Εδώ έχουμε και μια ταινία, ένα βίντεο σχετικά, Planet Within λέγεται. Είναι τρομακτική η εικόνα, δείχνει 40.000 τόνου ε, αποβλήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου δρόμου τη Ινδία και ανθρώπου με γυμνά χέρια να πιάνουν σκόνε και ένα σωρό επικίνδυνε χημικέ ουσίε ε, που καταστρέφουν την υγεία τους. Τα ηλεκτρονικά λοιπόν απόβλητα και ε, για μας και είναι πολύ ακριβή η επεξεργασία τους μεν, αλλά πρέπει να δούμε τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε για να τα διαχειριζόμαστε και επίσης τι οικονομικά κίνητρα στις αναπτυσσόμενες χώρες για τις εξαγωγές τους. Θα πρέπει ενδεχομένω να αποφύγουμε τη μεταφορά του ή να δημιουργήσουμε συνθήκε ασφαλού ε, επεξεργασία των ε, προϊόντων αυτών βλέπουμε ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται εδώς, εντός Ευρώπης μεν, αλλά δεν ανακυκλώνονται. Κάπου λοιπόν θα καταλήξουν αναγκαστικά. Εάν σκεφτούμε την παράνομη τώρα μεταφορά αποβλήτων, υπάρχει στρέβλωση στην αγορά αυτό και πλήττει και τους εμποροδόμενους και τους παραγωγούς και βλέπουμε αυτή είναι μια τάση αυξητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώ θα εντατικοποιήσουμε και θα εναρμονίσουμε τι διαδικασίε επιθεώρηση και ελέγχων. Αλλά θέλουμε και μια ευρωπαϊκή επισκόπηση για τι πηγέ ε, των αποβλήτων, το πώ συσχετίζονται αυτέ με άλλε παράνομε δραστηριότητε τη ε, συγκεκριμένη μετακίνηση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι είναι αυτό που επικοινωνεί αυτά τα φαινόμενα και πώ μπορούμε να τα αναχαιτήσουμε. Πώ μπορούμε να αναχαιτήσουμε την παράνομη μετακίνηση αποβλήτων και τι παράνομε εξαγωγέ του. Τέλο, η πληροφόρηση. Πάντοτε υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την συλλογή των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων. Το επαναλαμβάνω κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Το κόστο είναι ένα στοιχείο εδώ. Θα το δείτε όμω στην έκθεση μπροστά σα. ειναι αθαρρυντικό ενθαρρυντικό αυτό. Ότι κάποια κράτη-μέλη σε κάποιο επίπεδο έχουν την απέτηση να συγκεντρώνουν στοιχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα και τι διασυνοριακέ ε, μεταφορέ του με το πολύπλοκο σύστημα τη Σύμβαση τη Βασιλεία. Οι εξαγωγή όμω άλλων αποβλητών πρέπει να δίνουν πολύ λεπτομερέστε πληροφορίε για τι χώρε προορισμού. Όμω, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, υπάρχουν χώρε με πολύ λεπτομερέστερα στοιχεία. Θα μπορούσαμε και εμεί να συλλέγουμε λοιπόν περισσότερα δεδομένα χωρί πρόσθετε προσπάθειε. Θα πρέπει να ασκηθεί πίεση ώστε να υπάρχει τακτική υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση των, των ευρωπαϊκών δεδομένων με συγκεκριμένου ε, καταλόγου Εμπνεώμενοι από την περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων. Θα πρέπει να δούμε την υλοποίηση τη νομοθεσία και το κατά πόσο αυτή είναι ε, αποτελεσματική. Για το εμπόριο στα επικίνδυνα απόβλητα είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αλλά πρέπει να μετακινηθούμε από την διάθεση στην ανάκτηση και την ανακύκλωση. Και βεβαίω να αποφύγουμε την αναβολή των προβλημάτων μα αλλού. Το γεγονό ότι δεν συλλέγουμε τα αποβλητά αυτά ώστε να αξιοποιηθούν στη δική μα οικονομία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Γι' αυτό καταλήγουμε στο χαμηλό ποσοστό του 4%. Δεν είναι ότι δεν καταβάλουν προσπάθειες εταιρείε, απλώς κάποιες παράμετροι που λειτουργούν ταυτόχρονα ε, κάνουν αδύνατο το να μπορέσει κανείς να αντλήσει από κάποιο όφελος. Πάντως παραμένει γεγονό ότι εάν υλοποιήσουμε σωστά, καλύτερα μάλλον τι οδηγίε για τα επικίνδυνα απόβλητα, θα ανακτήσουμε ένα μέρος ανακυκλώσιμων. Θα δημιουργήσουμε ζήτηση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τη δική μα ζήτηση για πόρου. Είναι λοιπόν περίπλοκη η όλη αλυσίδα, αλλά δεν είναι αδύνατον ε, και εκτό κοινή λογική να σκεφτούμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Οι τεχνολογίε, τα επιχειρηματικά μοντέλα για λιγότερα απόβλητα ε, ή τουλάχιστον λιγότερο κίνδυνα απόβλητα, σχετικέ εγκαταστάσει, όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον περίπλοκο συσχετισμό μεταξύ των οδηγιών για τα απόβλητα και των συνεπειών όταν προσπαθούμε να δούμε και την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την ανάκτηση και την ανακύκλωση. Σχολίασα νομίζω και την ε, έκθεση που είχαμε μπροστά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Μακλέιντ. Η κυρία Τουτσίνσκα τώρα. του δικτύου Impel. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από τη δική μου πλευρά σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και με μεγάλη μας χαρά μοιραζόμαστε τα πορίσματα των εργασιών μας που είμαστε το Impel, δηλαδή είμαστε ένα δίκτυο που παρακολουθεί την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Έχουμε 46 μέλη που προέρχονται από 33 χώρες. Δεν είμαστε λοιπόν μόνο χώρες μέλη, δεν είμαστε καν χώρες μέλη, είμαστε ε, οργανώσεις οι οποίες εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε θελοντική βάση γιατί νομίζουμε ότι αυτό προσφέρει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια ε, των αρμόδιων και υπεύθυνων ε, περιβαλλοντικών αρχών. Υπάρχουμε από το 1992 20 χρόνια λοιπόν συμπληρωμένα φέτος και τα θέματα αυτά που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξή σας σήμερα αποτελούν μέρος και του δικού μας προγράμματος εργασιών τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μάλιστα νομίζω θα φανεί, θα αποδειχθεί ότι είναι και προτεραιότητα για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι το 2015. Λέγομαι λοιπόν Σοφία Τουτσίνσκα, ε, είμαι Σουηδή και πρόεδρος του ΙΜΠΕΛ Έχω κοντά μου δύο σημαντικά πρόσωπα, την Μάγδα Γκόσκ από το Σουηδικό Chief Inspectorate, την ε, Επιτροπή που παρακολουθεί τις ε, μεταφορές και για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, για τα προγράμματα δηλαδή επιβολής, εφαρμογής και κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την εξέταση των μεταφορών, αν δηλαδή η κάθε συγκεκριμένη μεταφορά είναι σύμμορφη με τις διατάξεις. Θα συζητήσουμε, δεν θα συζητήσουμε τόσο πολύ αν ε, γίνονται μεταφορές υπερβολικά προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά ε, ο βασικός μας καθήκον είναι να είμαστε επιτόπου και να εξετάζουμε και διαπιστώνουμε ότι γίνονται σωστά οι μεταφορές. Επίσης, πολύ σύντομα θα προσκαλέσω τον project manager να σας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με το έργο μας, ποια είναι δηλαδή το συνεχιζόμενο έργο μας. Έχω πρώτα να σας πω λίγα γενικά συμπεράσματα ε, από την εργασία μας. Μεταφορές αποβλήτων και διαμεθοριακά. Έχουμε κάνει μια σειρά project από τις αρχές του 2000 και συνεχίζουμε ποιο είναι το περιεχόμενο και με ποιο τρόπο γίνονται. Εμείς συνερχόμαστε, συμφωνούμε για κάποια προγράμματα επιθεωρήσεων καθώς και το χρονοδιάγραμμα και μετά προχωρούμε στη συλλογή των δεδομένων. Το 2012 έγιναν πάνω από 8.000 επιθεωρήσεις μέσα στα πλαίσια της οργάνωσής μας και για μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για μεταφορές οι οποίες διαβαίνουν τα σύνορα της Ένωσης. ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που προκύπτουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε από τις επιθεωρήσεις μας ότι οι παραβιάσεις των ισχυουσών διατάξεων βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο όπως την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε ας πούμε ένα ρυθμό παραβιάσεων της τάξης του 20%. 20% λοιπόν των επιθεωρήσεων ενετόπισαν κάποιο είδος παραβιάσεως ε, των κανόνων που ισχύουν για τις μεταφορές. Μπορούν να διαφοροποιηθούν οι παραβιάσεις αυτές, να χωριστούν σε δύο ομάδες, μία που έχει περισσότερο σχέση με τις εσωτερικές, τις ενδοενωσιακές μεταφορές, όπου ε, είναι ας πούμε ελλειπή τα έγγραφα, δεν έχουν τις ε, σωστές ημερομηνίες ή τα σωστά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, μεταφορές εκτός ενώσεως, είναι προς χώρες μη όσα που ε, απαγορεύεται η εξαγωγή, τους, η εξαγωγή των απορριμμάτων, δηλαδή των αποβλήτων, στις χώρες αυτές. Ηλεκτρικά, ε, ηλεκτρονικά είδη και οχήματα που έχουν, ε, έχει λήξει πλέον ο κύκλος ζωής τους. Καμιά φορά αυτά αναφέρονται ως ήδη ως αγαθά τα οποία μπορεί, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Από τις μεταφορές αυτές, για να είμαι πιο συγκεκριμένες, 41% ε, ανασχέθηκαν, σταμάτησαν, διακόπηκαν. Υπήρξε και ένας αριθμός που επανήλθαν, επιστράφηκαν δηλαδή στον ε, Αποστολέα. Ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τις δραστηριότητες αυτές και τι επιζητούμε με το συνεχιζόμενο έργο μας. Εμείς πιστεύουμε πρώτα ότι το γεγονό και μόνο ότι συνεργαζόμαστε, τα μέλη δηλαδή, ενθαρρύνουμε τον τρόπο αυτό την εκτέλεση επιθεωρήσεων. Αυτό ήδη σημαίνει προστιθέμενη αξία. Βέβαια γίνονται πολύ περισσότερες επιθεωρήσεις και έλεγχοι και εκτός, από τις, εκτός του πλαισιού μας δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές. Αλλά είναι μια συστηματική κοινή προσπάθεια και εξακολουθεί για μας να είναι προτεραιότητα. Κάτι το οποίο επίσης αποτελεί ε, κέριο χαρακτηριστικό και ίσως δεν έχει συζητηθεί ακόμη, είναι η ανάγκη συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες αρχές, όπως εισαγγελικέ αρχές, αστυνομικές, λιμενικές αρχές. Χωρίς καλή και στενή συνεργασία, η αλυσίδα των επιθεωρήσεων θα σπάσει, αν δεν μπορούμε δηλαδή να συνεργαστούμε στενά. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά με τις αρμόδιες αυτές αρχές για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων μας. Ένα άλλο στοιχείο που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την βελτίωση των αποδοτικό, της αποδοτικότητάς μας είναι να πάμε και προς τα ανάντι, δηλαδή όχι μόνο τις μεταφορές που βρίσκονται ή στο δρόμο ή στο λιμάνι, αλλά να δούμε από πού προέρχεται η μεταφορά, από πού προέρχεται το απόβλητο. Το τελευταίο που έχουμε στην ατζέντα μας είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια εντατικοποίησης της συνεργασίας με τις χώρες και με τις περιβαλλοντικές αρχές που δέχονται στα εδάφη τους, στις επικρατείες τους αμφισβητούμενα απόβλητα. Για παράδειγμα με χώρες της Δυτικής Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και αυτά για μας είναι ε, κρίσιμα πράγματα για να είμαστε πιο επιτυχείς στην αντιμετώπιση των παράνομων αυτών μεταφορών. Βλέπουμε ακόμη και το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι κοινέ μας αυτές οι συνεργασίες, αλλά είμαστε πιεσμένοι κάπως από ψηπόρων. Έχουμε περιορισμούς. Έχουμε επίσης τώρα εκθέσεις από παλαιότερες παλαιότερες ε, εργασίες μας που είναι στην ιστοσελίδα μας impel.eu και αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος ε, να παρακαλέσω να δοθεί ο λόγος στον Project Manager να σας δώσει λίγες λεπτομέρειες για, για το έργο κοινών επιθεωρήσεων που διεξάγεται ε, τώρα. Ευχαριστώ. Κέιτι όλοι. Όπως είπε η Σοφία, ε, το πρόγραμμα αυτό μας, δίνει τις, ε, μας δείχνει τις ε, δραστηριότητες εφαρμογής τις εννέας μέρες, εννέας μέρε, εννέα μέρες συγγνώμη, επιθεωρήσεων που κάναμε, είδαμε μια εικόνα. Έχουμε αποτελέσματα από 23 χώρες και καλύψαμε πολλές χιλιάδες ε, αποστολές αποβλήτων και 110 εταιρείε. Το 67% των ε, επιθεωρήσεων ε, έγιναν επιτόπου. Είχαμε ποσοστό παραβιάσεων 21%. 29% ήταν το ποσοστό παραβιάσεων της εταιρεία. Επομένως, θα πρέπει πολύ νωρίς να ανοιχνεύσουμε τα προβλήματα. 1.120 περίπου επιθεωρήσεις Είχαμε και πληροφορίες αυτές. 1.500 τις επιλέξαμε και οι υπόλοιπες ήταν τυχές. Ε, είχαμε ε, απόβλητα ηλεκτρονικά και οχήματα στο τέλος ζωής τους, ελαστικά, εκεί ήταν οι περισσότερες παραβιάσεις. Οι χώρες προορισμού ήταν 39% των παραβιάσεων ήταν χώρες εκτός ΩΣΑ, ε, Η Κίνα κυρίως ήταν ο πιο συχνός προορισμός. Εν συνεχεία, τι κάναμε μετά από τις επιθεωρήσεις, 91%, ε, ε, συγγνώμη, επαναπατρισμούς, 89 κυρώσεις, 56 προειδοποίησεις και μερικές δεκάδες, 13 διώξεις. 5.500 ε, είχα, επιθεωρήσει είχαμε με ε, τη βοήθεια τελωνιακών αστυνομικών και 3.800 ε, με τη βοήθεια άλλων αρχών. Δεν έχουμε ακόμα αναλύσει τα δεδομένα λεπτομερώς. Εξακολουθούν να έρχονται για φέτος από τις πληροφορίες. Όταν είχαμε επιθεωρήσεις με συνοδεία πληροφοριών, είχαμε εντοπίσαμε περισσότερα προβλήματα. Βέβαια και οι τυχαίες επιθεωρήσεις είναι σημαντικές για να δούμε το επίπεδο μη συμμόρφωση. Ευχαριστώ. Νομίζω ακούσαμε τις παρουσιάσεις. Κατέστη σαφές. Ότι εδώ εξάγονται εκτός των συνόρων και πρώτες ύλες και υπάρχει μια δυνατότητα σημαντική, εάν τα σταματήσουμε αυτά, να επιτύχουμε κάτι και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και 400.000 θέσεις απασχολήσεως στην Ευρώπη, εάν μπει φρένο σε αυτές τις παράνομες εξαγωγές. Έτσι λοιπόν το θέμα πρέπει να προσεγγιστεί από διάφορες πλευρές και από την σκοπιά των πρώτων υλών, της βιομηχανικής πολιτικής, πολιτικής περιβάλλοντος, αλλά και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια δημιουργίας απασχόλησης. Βέβαια, έχω ορισμένους συγκεκριμένους συναδέλφους και πρώτος είναι ο Βιτόριο Πρώτη και μετά θα ακολουθήσει η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Καλώς ορίσατε και εσείς ως πρώτη χριστιανοδημοκράτησα εδώ την παρέα μας σε, ως τέταρτη θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη Ριάγια Μαγκλέιντ και τους συντάκτες της έκθεσης. Για να ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις του Πρόεδρου μας, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει βιομηχανική πολιτική και έχει συγκεκριμένη έκφραση ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε σε μια συγκέντρωση με μεγάλη προσέλευση μηχάνων της Ευρώπης και αυτά έπαιγε σε ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια προσέγγιση συνεπή, συνεκτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς και αυτές οι μεταφορές αποβλήτων αυτό δείχνουν ότι πόρους έχουμε, αλλά θα πρέπει να μας οδηγήσουν. Μάλλον θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές, σαν να είναι πραγματικοί πόροι. Συνοψίζοντας λοιπόν, από το 2000 έως το 2009 βάσει της έκθεσης, αυξήθηκε κατά 28% η μετακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων επίσης αυξήθηκε κατά 131%. 2,42 ε, εκατομμύρια τόνους. Η εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από χώρες εκτός Ένωσης αυξήθηκε κατά 197% και η παραγωγή αποβλήτων που εξήχθησαν για για διάλυση έφτασε το 20, 27, αυξήθηκε κατά 20-27%. Η ανταλλαγή των ε, παράνομων ηλεκτρονικών αποβλήτων συνεχίζει όπως ε, επισημάνθηκε. ο Οργανισμός για το Περιβάλλον ε, υπολόγισε για το λιμάνι του Αμβούργου μόνο ότι μετακινήθηκαν τουλάχιστον 93.000 τόνοι προς την Αφρική, προς τη Δυτική Αφρική. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αύξηση των διασυνοριακών μεταφορών των αποβλήτων. Θα μπορούσε να μας πει ο υπεύθυνη του οργανισμού περιπολόντος και ποιο λόγο υπάρχει τέτοια έκρηξη στην μετακίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων σίγουρα Υπάρχει διαφορά στην, στο κόστος επεξεργασίας. Όπως λέγεται και στο κείμενο, οι τιμές αντιμετωπίζονται ως το βασικότερο κίνητρο από τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων και πλαστικών, μεταλλικών, χάρτινων, αυτά εξάγονται συνήθως προς την Ασία σε όγκο και τιμή ανάλογο των εξαγωγών που έχουν φτάσει υπέρμετρα ε, μεγέθη. Το 2011 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τους 18 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, μετάλλων και χάλιβα με αξία 7 δις ευρώ, με 12 εκατομμύρια τόνους χαρτιού, αξίας 1,6 δις ευρώ και 4 εκατομμύρια τόνους πλαστικού με αξία 1 δις ευρώ. Αυτό λοιπόν που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι, μην ξεχνάμε και τη χθεσινή πρόταση που είδαμε, τη διάλυση των σκαφών. Ε, υπάρχει εδώ δυνατότητα εφαρμογής του πρωτοκόλου της Βασιλείας και θα μπορούσαμε έτσι να σπρώξουμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπουμε πώς ε, αντιμετωπίζεται η διάλυση των σκαφών αλλού τι θα πει αλλού. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, παραμελούμε τους πόρους μας. Προς όφελος του περιβάλλοντος και του δικού μας θα μπορούσαν αυτοί οι πόροι να μένουν στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να διεξαγάγει από αυτή την έκθεση είναι δυστυχώς ε, λυπηρά. Α, μετά από 30 ετή, 30 ετή, εφαρμογή τη οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα, βλέπουμε να μην υπάρχει φιλική προ το περιβάλλον επεξεργασία των αποβλήτων και να παραβιάζονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι εξαγωγέ των επικίνδυνων αποβλήτων συνεχώ αυξάνονται. Η παράνομη μετακίνηση αποβλήτων επίση αυξάνεται, ιδίω ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Και ο ΙΕ και η Ιντερπολ δήλωσαν ότι οι μετακινήσει αυτέ ουσιαστικά έχουν πλέον περάσει στα χέρια των ε, οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Αυτό είναι ένα σημαντικό πόρισμα της έκθεσης αυτής. Η όλη δραστηριότητα των αποβλήτων, της μεταφοράς αποβλήτων, επιτρέπει και τη λεύκανση παράνομων προσόδων από τις παράνομες εγκληματικές ομάδες. Εδώ βλέπουμε με την έκρηξη των εξαγωγών ε, μετάλλων, πολύτιμων μετάλλων, χάλιβα, ε, σιδήρου, νικελίου, χαρτιού, πλαστικού προς την Ασία, βλέπουμε ότι αυτό ουσιαστικά ε, φέρει, αποφέρει κέρδη σε ένα περιορισμένο αριθμό εμπορευομένων και αποστερεί την Ευρώπη από σημαντική πόρους μετάλλων και ενέργειας. Η δυνατότητα να συλλέξουμε στοιχεία και να τα εξετάσουμε με προσοχή για την εξαγωγή των αποβλήτων είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατεπηγόντω. Για να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση και την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά και μη επικίνδυνων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ίσω ένας οργανισμός ή έστω μια θέση εντό του υπάρχοντος οργανισμού όπου θα συγκεντρώνονται σε κεντρικό επίπεδο τα ε, δεδομένα για τα απόβλητα και τις ε, μεταφορές τους και να δημιουργεί σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, τις ροές οικονομικές και προϊόντων ώστε να μην δημιουργείται μια αγορά αδιαφανής που αφήνει περιθώρια για ε, παράνομες δραστηριότητες. Θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία για να έχουμε ωφέλη για τα κράτη-μέλη και επίσης να δημιουργηθούν κοινοί μηχανισμοί ώστε να παρακολουθούμε τις μετακινήσεις των αποβλήτων. Σύλλογα για 14 έχουμε ένα χάρτη. Ε, μια περίπτωση στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Βιτόριο. Λίντα Μακάβαν. Ξέρω από το δικό μας οργανισμό περιβάλλοντος ότι οι εξαγωγές κυρίως ηλεκτρονικού υλικού είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχουν και πρώην αξιωματικούς της αστυνομία που συνεργάζονται μαζί τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα, φαίνεται πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με την ανακύκλωση Με ποιο τρόπο γίνονται οι έλεγχοι ώστε πραγματικά να γίνεται η πραγματική ανακύκλωση. Ε, υπάρχει υποχρέωση να δημοσιεύει κανείς πού πάνε τα πράγματα που ανακυκλώνει. Γιατί διότι εδώ κάποιοι νύπτουν τα σχήρα τους, δηλαδή τα πουλάνε και τα ξαναπουλάνε και παραπέρα τα πουλάνε. Είχαμε χθε και τη συζήτηση για την αυσιπλοεία, για την ναυτιλία. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι το ίδιο. Δηλαδή το καράβι το πουλάει ο πλειοκτήτης έναν παραπέρα και αυτός παραπέρα και αυτός παραπέρα και κάπου χάνονται τα του. Και ο κόσμος ανησυχεί. Μου στέλνουν γράμματα. Κάνουν ε, όλο αυτό το μπελά, δηλαδή περνάνε όλοι αυτοί, όλο αυτό το μπελά, κάνουν αυτή προσπάθεια να χωρίζουν τα ε, οικιακά τους απορρίμματα και μετά βλέπουν ε, εικόνες, ε, φωτογραφίες παιδιών στον Μπαγκλαντές τα οποία διαλύουν ε, παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λένε «Μα τι γίνεται». Λοιπόν, το πρόβλημα πού βρίσκεται. Υπάρχει πράγματι πολιτική βούληση στις χώρες μέλη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μήπως οι δημόσιες αρχές πρέπει να εξηγήσουν, να δημοσιεύσουν, να, δηλώσουν δημοσία δηλαδή πού πάνε τα ανακυκλωμένα αγαθά. Ευχαριστώ. Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι παρούσες και παρόντε. Βέβαια, η πέμπτη απόγευμα δεν είναι και ιδεώδε χρονικό διάστημα. Τώρα, πρώτο ερώτημα είναι, αρκούν οι έλεγχοι. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερα πράγματα εάν είχατε περισσότερους πόρους. Τώρα, έλεγχος αλλά έλεγχος πάνω σε τι. Ήδη ο ορισμός του απορρίμματο ή αποβλήτου μπορεί να ερμηνευτεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Για το εμπόριο Χρειάζονται βεβαίω πάντοτε δύο. Ένας ο οποίος στέλνει και ένας ο οποίος δέχεται. Από τη στιγμή που το απόρριμα δεν είναι σκουπίδι αλλά είναι εμπόρευμα, πού θα κάνετε την επαλήθευση, πού θα κάνετε τον έλεγχο. Δεν θέλω να με παρανοήσετε, εγώ είμαι αντίθετη με οποιαδήποτε αποστολή, με οποιαδήποτε μεταφορά απορριμμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σαφέστατες ρυθμίσεις ούτε θέλουμε τις βρωμιές μας να τις στέλνουμε έξω. Αλλά ξαναθέτω το ερώτημα. Πώς ορίζονται, δεν αρκούν βεβαίως οι έλεγχοι μόνο των εγγράφων, διότι το έγγραφο, όπως λένε, το χαρτί, είναι υπομονητικό. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και επί τόπου Και το ερώτημα επίσης είναι, από πού θα βρείτε υποστήριξη. Έχετε υποστήριξη των ντόπιων αρχών στα λιμάνια υποδοχής και ε, σε, στις επιχειρήσεις που δέχονται τα απορρίμματα ε, ή απόβλητα. Ε, βλέπω λοιπόν να θιθεται πολλά ερωτήματα στον χώρο αυτό. Εν τέλει, οι εμπειρογνωμόνων μας για ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρονικά απόβλητα δηλαδή, η κυρία Βαν Μπρέμπτ Χαίρομαι που με συγκαταλέγεται μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Δεν είμαι πραγματική εμπειρογνωμόνων, ωστόσο με παθιάζει το θέμα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία μας υποβάλλατε. πολύ ίδιοι, πολύ ήδη είπαν ότι είναι παράξενο, ενώ χρειαζόμαστε τα υλικά αυτά και ιδίω τις πρώτες ύλε που προκύπτουν από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών. Η οικονομία μας τα χρειάζεται αυτά. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρει αυτό το λάθος δρόμο των παράνομων εξαγωγών και δεν καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Ε, επανεπεξεργαστήκαμε την οδηγία προσφάτως και προσπαθήσαμε εμείς να περάσουμε τις θέσεις μας και απέναντι στο Συμβούλιο που Εμείς δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε ακόμα πιο έντονους τους ελέγχους, πιο δύσκολες τις εξαγωγές αυτές. Αυτή η νέα οδηγία καλύτερο πλαίσιο ή ε, θεωρείτε ότι είναι καλύτερο πλαίσιο ή χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλειών διότι εξετάζοντας τα αριθμητικά στοιχεία ε, είναι πραγματικά ανισχυτικά. Η αγορά χρειάζεται τις πρώτες ύλε που προέρχονται από τα απορρίμματα αυτά. Και όμως χάνονται. Δεύτερο, εγώ είμαι από την, προέρχομαι από την Αμβέρσα και είναι γνωστό το λιμάνι της Αμβέρσας, πιθανώς και σε εσά. Για ένα διάστημα μάλιστα εργάστηκα και ε, στην ε, διοίκηση του λιμανιού της Αμβέρσας και γνωρίζω τις προσπάθειες που γίνονται εκεί να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι παράνομε εξαγωγέ ηλεκτρονικού υλικού. Αλλά και στη δική σας χώρα κύριε Πρόεδρε υπάρχουν σχετικά παραδείγματα διότι γίνονται και εισαγωγέ αποβλήτων και μάλιστα όχι ασήμαντες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι στις εισαγωγές αυτές περί τίνος κυρίως πρόκειται. Είναι πάλι εκεί ηλεκτρονικό υλικό ή είναι άλλο υλικό. Και τελικώς που καταλήγει, τι γίνεται. Είναι αρκετά αυστηρή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Η Κομισιόν πρώτη. So, um... Uh, uh, mm, uh, Ο κύριος Πρόντι έκανε κάποια σχόλια και έθεσε πολυπίκυλα θέματα. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Μας απασχολούν οι εξαγωγές πολύτιμων αγαθών ή πολύτιμα απόβλητα, αν θέλετε, σε τρίτες χώρες. Έχουμε μια προτεραιότητα αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων. Ε, έχουμε μια πολιτική αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων. Είναι κακό για την οικονομία, είναι κακό για το περιβάλλον κάτι τέτοιο. Και εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Πρώτον, οι εξαγωγές πολύτιμων αποβλήτων είναι ένα τμήμα του προβλήματος μόνο. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τα βέλτιστα. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες στατιστικές για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσίευσε η Eurostat το Μάρτιο του 2012. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. δείχνουν ότι για τα αστικά απόβλητα οι χωματερές είναι η κυριότερη λύση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 50% όλων των αστικών αποβλήτων καταλήγουν σε χωματερές. Με βάση τα σημερινά συστήματα λοιπόν, αντί να χρησιμοποιούμε αυτά τα απόβλητα ως ε, πόρους, απλώς θα θάβουμε σε τρύπες. Θα θάβουμε σε χωματερές. Δημοσιεύθηκε και ένας πίνακας ε, επιδόσεων και αποτελεσμάτων τον Αύγουστο για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Και με, με ενδιαφέρον μπορούμε να δούμε ότι πάνω από 10 κράτη-μέλη έχουν ποσοστά χρήσης της χωματερής για τα αστικά απόβλητα πάνω από το 75%. Όλα τα οικιακά απόβλητα, όλα τα αστικά απόβλητα, το 75% αυτών, καταλήγουν σε χωματαρίες. Κάτι το οποίο είναι κατά της πολιτικής μας ε, για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Για τα επικίνδυνα απόβλητα τώρα. Οι μετακινήσεις ε, επικίνδυνων αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι το βασικό μας πρόβλημα. Και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες εκθέσεις δείχνουν ότι γίνονται αποστολές επικίνδυνων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και για να χειριστούμε αυτά τα απόβλητα θέλουμε πολύ εξελιγμένες εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και για να κάνουμε μία βέλτιστη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, χρειαζόμαστε αυτή τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα υπάρχει μια άλλη πτυχή που πραγματικά είναι ανησυχητική. Η παράνομη απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στα κράτη-μέλη. Συμβαίνει αυτό, είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου οι ροές επικίνδυνων αποβλήτων παρακολουθούνται, αλλά καθημερινά λαμβάνουμε αναφορές και παράπονα που δείχνουν ότι αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται παράνομα στα κράτη-μέλη. Το ερώτημα της κυρίας Μακάβαν. Μία βασική προϋπόθεση για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κάνουμε μεγαλύτερο διαχωρισμό στη συλλογή των αποβλήτων. Είναι καλύτερη λύση από περιβαλλοντική σκοπιά. Και μας δίνει μια καλή βάση για να προωθήσουμε το σύστημα της ανακύκλωσης. Υπάρχει αυτό στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα το ερώτημα της κυρίας Κλάς. Υπάρχει συνένεση ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους είναι τα κύρια μελήματά μας. Είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Η κυρία Βαν Μπρένταν μα, μας ρώτησε αν αρκεί η αναθεώρηση. Ναι, νομίζουμε. Αυτή η αντιστροφή του βάρους απόδειξης πιστεύουμε ότι θα είναι δυνητικά χρήσιμο εργαλείο. Όλα εξαρτώνται από το πώς η οδηγία αυτή η αναθεωρητική θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Κομισιόν θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές, κατευθύνσεις γενικά για την ερμηνεία και εφαρμογή της νέας αυτής οδηγίας. Θα το έχουμε υπόψη μας αυτό το θέμα. Και θα δούμε πώς την εφαρμόζουν οδηγία αυτή τα κράτη-μέλη. τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους. Εδώ σαν υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Ο αριθμός αυτών των οχημάτων ο αριθμός αυτών των οχημάτων που αναφέρει η Eurostat ότι δεν ξέρουμε που καταλήγουν είναι τεράστιος η εξαγωγή αυτοκινήτων παλιοσίδερων είναι σημαντικό θέμα, σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση των εξαγωγών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Αυτό το μέσο δεν είναι υποχρεωτικό. Όταν δημοσιεύσαμε το πρόγραμμα της Κομισιόν, θα κάνουμε έναν έλεγχο καταλληλότητας κάποιων νομοθετημάτων και η σχετική οδηγία θα αξιολογηθεί. Και ο έλεγχος καταλληλότητας θα γίνει ούτω ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο κενό στην εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Επιθυμεί κανείς άλλος. Α, η κυρία Τουτσίνσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Από τη σκοπιά της Ίμπελ. οι ερωτήσεις σας αναφέρονται και στην πολιτική αλλά και στην εφαρμογή της ισχύουσας πολιτικής και νομοθεσίας και που βρισκόμαστε τώρα. Θα ήθελα να στοχεύσω τα σχόλιά μου και τις απαντήσεις στα θέματα της εφαρμογής που είναι και ο βασικός όγκος των καθηκόντων της ΙΜΠΕΛ Έχουμε την νομοθεσία, ναι, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Η απάντηση είναι ναι. Και τα μέλη μας, περιβαλλοντικές αρχές, εργάζονται σκληρά και αναλαμβάνουν τις απαραίτητες δράσεις. Είμαι βέβαια ότι μπορούν να βρεθούν τρόποι βελτιώσεως και αυτή είναι και η προσπάθειά μας. Υπάρχουν και οικονομικές δραστηριότητες που δεν είναι καταρχήν παράνομες. Είναι όμως πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις οικίες περιβαλλοντικές αρχές. Όπως έχουμε διαπιστώσει από τις επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις άλλες υπεύθυνε ρυθμιστικές αρχές και να δούμε επίσης που είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα καθήκοντα αυτά στα πλαίσια αυτών των αρμόδιων αρχών, όπου δηλαδή η μεταφορά ε, αποβλήτων δεν είναι η πρώτη στη ε, προτεραιότητά τους. Για να βελτιωθεί η κατάσταση νομίζω πρέπει να διατηρούμε στενότερες επαφές με τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρες εκείνες που είναι οι χώρες υποδοχής των αποβλήτων και μεγάλου μέρους βέβαια των παράνομων αποβλήτων ή απορριμμάτων. Έχουμε την ε, Σύμβαση της Γενέβης που μας δίνει τα εργαλεία αλλά και σε αυτές τις αρχές να παίξουν τον σωστό ρόλο των εταίρων μας για την διασφάλιση της ορθότητας των μεταφορών και οι εταίροι μας στη Νοτιοανατολική Ασία ή Δυτική Αφρική είναι ασθενείς, είναι αδύναμοι και χρειάζονται από μας συνεργασία μέσω δικτύων για να βελτιωθεί η ικανότητά τους να εφαρμόσουν ε, από τη δική τους πλευρά τα προβλεπόμενα. Τέλος, νομίζω ότι κάναμε πρόοδο Έχουμε βελτιώσει το έργο των περιβαλλοντικών αρχών. Έχουμε πάντως καλύτερα μέσα στη διάθεσή μας τώρα με, τον την αναθεωρημένη οδηγία, για παράδειγμα και για μεταφορές που υποπτευόμαστε ότι είναι ε, παρανόμως επισημασμένα ως ε, φορτία, δηλαδή τα οποία είναι παρανόμως επισημασμένα ως ε, ε, υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ευχαριστώ κύριε Μαγκλέιντ. Σα ευχαριστώ να απαντήσω σε μερικέ από τι συγκεκριμένε παρατηρήσει για την έκθεση και μετά να κάνω κάποιε γενικότερε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το μεγάλο βέλο κατευθύνεται προ τη Γερμανία, γιατί υπάρχουν καλύτερε εγκαταστάσει, προηγουμένες τεχνολογίε και μέσα τεράστια δυνατότητα δηλαδή. Και τα σύνορα είναι κοινά με πολλέ χώρε. Οπότε πολλοί στέλνουν προ τη Γερμανία. Αυτό είναι ο βασικό λόγο. Όμω αυτό αλλάζει το γεγονό ότι στα πλαίσια τη βιομηχανική πολιτική υπάρχουν τεράστιε αποκλήσει μεταξύ των χωρών. Και το θέμα είναι ακριβώς πώς θα γίνει αυτός ο συνδυασμός, διότι εάν ε, υπάρχει κάποια αξία στην αγορά εδώ και αν δείτε στην έκθεση της σελίδα 23 θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σοβαρές ε, δυνατότητες ε, να αποκομίσουμε αξία χάρη στη μετακίνηση των αποβλήτων. Όμως δεν συνειδητοποιούμε την πραγματική αξία των αποβλήτων και αυτό είναι το πρόβλημα. Η συζήτηση είναι... Δεν έχει δώσει λύση για τις τιμές ενέργειας λόγω χάρη, την αποτέφρωση που θα την ενέργεια θα μπορούσε να προκύψει από την αποτέφρωση. Τι σύγκριση μπορεί να γίνει με την ε, αγορά που, με την τιμή που προκύπτει στην αγορά αποβλήτων. Δεν ξέρω λοιπόν εάν ο συσχετισμός, αυτός ο πολλαπλό συνδυασμό μπορεί να δώσει πραγματικά κινήτρα για την αγορά. Συμφορώ πάντως μαζί σας ότι πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση εδώ. Διότι πραγματικά το πιο απογοητευτικό είναι να βλέπει κανεί να μπαίνουν όλα σε ένα φορτηγό και να φεύγουν προ έχουν στην κατεύθυνση. Ε, Πάντω, ναι, στη Δανία βλέπουμε να περνάνε φορτηγά και να ζητάνε οτιδήποτε υπάρχει σε απόρριμα απόβλητο για να το κάψουν στο το πιο γρήγορα. Βλέπουμε πόσο γρήγορα έχει προχωρήσει εκεί η υποτέφρωση. Πάντω, το γεγονό ότι η σύμβαση τη Βασιλεία δεν έχει συγκεκριμένο συγκεκριμένη πρόβλεψη γι' αυτό σε επίπεδο του οργανισμού περιβάλλοντος. Επιβάλλει ένα είδος ε, καταλόγου κωδικών για τα κράτη-μέλη και την υποβολή εκθέσεων. Βεβαίω, θα είναι πολύ πιο έτοιμοι όσοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς αυτούς να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίε για τον WE. Εάν δείτε τους αριθμούς θα δείτε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και το τι αριθμοί καταγράφονται τελικά στις, ε, στη Γερμανία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά που τα αποθηκεύουν σε υπόγεια, σε σοφίτες και το καθεξής. Όμως, είναι πολλέ τηλεοπτικέ συσκευέ, οι παλιέ τηλεοπτικέ συσκευέ που πηγαίνουν προ την Αφρική λόγω χάρη. Ξέρουμε ότι δεν θα λειτουργήσουν τελικά, δεν πρόκειται να χρησιμοποιούν, θα καταλήξουν στα σκουπίδια, σε ένα απόμερο μέρο τη πόλη ενώ κάποιοι θα χάνουν μεστούς και χάνεται και, και ενδεχόμενο κέρδος από αυτά τα απόβλητα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε το, το δυναμικό, ε, το οικονομικό που διαθέτουν τα απόβλητα. Καλωσορίζω λοιπόν τις επιθεωρήσεις που θα πρέπει να βασίζονται ακριβώς ε, σε ευφυή αναζήτηση, αλλά περισσότερη σημασία έχει ακόμη να έχουμε λεπτομερέστατες διεξοδικές εκθέσεις στην υποβολή τους θα μπορούσαμε έτσι να διαχειριστούμε το όλο θέμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Οι πληροφορίε θα μα βοηθήσουν ακριβώ να είμαστε πιο αποδοτικοί στο να εντοπίζουμε και να καταγράφουμε σωστά τι μετακινήσει. Τώρα για όσα είπε η κυρία Κλάς για τους ελέγχους. Ε, βλέπουμε ροή καλών πληροφοριών στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας να μας βοηθά πάντοτε τρομερά ε, και να βοηθούν την καλύτερη υλοποίηση τη οδηγία. Να ολοκληρώσω μια τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα, Βιτόριο. Η λεύκανση προσόδων και η απώλεια πόρων είναι πραγματικά κάτι που ε, χαρακτηρίζει την ε, επεξεργασία αποβλήτων. Η πηγή, ο προορισμός και η κωδικοποίησή τους θα ήταν πραγματικά ένα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι έκαναν τις παρουσιάσεις, έδωσαν απαντήσεις και έκαναν βεβαίω ερωτήσεις. Μας προσφέρατε σημαντική τροφή για σκέψη. Ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν και πολύτιμες πρώτες ύλες, τις οποίες χάνουμε. Άρα εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή, να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμεθα. Ευχαριστώ. werden einmal noch schnell umbauen. Genau. Und jetzt geht... Ευχαριστώ. Τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι το υπαριθμό 23 και αναφέρεται στη χρηματοδοτική κρίση στο Διεθνές Ταμείο για καταπολέμηση του AIDS, φυματίωσης και ελονοσίας και οι επιπτώσεις της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται ιδιαίτερως από την ελονοσία και που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε πολλαπλά φάρμακα, ιδίω δε στην Ρουμανία. Καλωσορίζω την, την εκπρόσωπο της Κομισιόν, καθώς και τον κύριο Μουσα, Μασούντ Νταρά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που έχει προσέλθει για να συζητήσει μαζί μας ε, το πολύ σημαντικό αυτό θέμα να διευκρινίσουμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα τεχνικά θέματα πρώτα. So everything is fine, everything is prepared. Dann können wir starten und Sie haben jetzt ausschließlich das Wort für die Präsentation. Λαμβάνετε το εσείς τώρα για να κάνετε την παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Εκ μέρου ε, ε, του Γραφείου για την περιοχή της Ευρώπης από τον ΠΟΗ και των συναδέλφων της Αντιπροσωπείας παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, θυματίωση και την ε, ανθεκτική σε πολλαπλή στην, ε, στα φάρμακα μορφή της θυματίωσης και το τι συμβαίνει στην περιοχή της Ευρώπης και παγκοσμίω. Μιλάμε για μια περιοχή με 53 κράτη-μέλη του ΠΟΗ και με ένα πληθυσμό των 900 εκατομμυρίων περίπου. Υπάρχει ένα ενοποιημένο πρόγραμμα για να αναχαιτήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την ε, θυματίωση αυτού του τύπου MDR-TB, ιδίω στη Ρουμανία. Θα δούμε τι βασικέ προκλήσει, μάλιστα, σε σχέση με τι μορφέ αυτή τη θυματίωση στην ε, περιοχή αυτή. Έχουμε 8,8 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίω στη θυματίωση. Αν δούμε τη γεωγραφική κατανομή, έτσι περίπου θα εμφανιζόταν όπως στο διάγραμμα ο παγκόσμιος χάρτης. Βλέπουμε να γίνονται πολύ μεγάλες η Αφρική και η Ασία και να μικραίνουν πάρα πολύ η Ευρώπη. 5% της πίεσης από τα κρούσματα θυματίσεως ασκούνται στην Ευρώπη. Όμως η μορφή της MDR ε, ε, είναι εκείνη που περισσότερο συναντάται στην Ευρώπη και είναι και πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι που μας πλήττει περισσότερο. Έχουμε 300, ε, κρούσματα ετησίως στην περιοχή της Ευρώπης, 81 περιπτώσεις που καταγράφονται, 80.000 περιπτώσεις που καταγράφονται και 45.000 θανάτους. Είναι πραγματικά πολύ παράξενο να σκεφτόμαστε ότι έχουμε θανάτους από την θυματίωση στην Ευρώπη ακόμη. Πάντως, υπήρξε μια μείωση από το 2005, αλλά είναι πολύ μικρή η μείωση αυτή, πολύ αργή. Δεν φτάνουμε τους στόχους της χιλιετίας όπως έχουν γνωριστεί στην όλη περιοχή. Έχουμε 53 κράτη-μέλη, όπω είπα. Τα 18 από αυτά ονομάζονται χώρες υψηλή προτεραιότητας. Είναι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επιπλέον η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Με πράσινο βλέπετε τις χώρες που και αυτές ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από που δεν έχει εκκριζωθεί η θυματίωση. Δεν αφορά λοιπόν μόνο τις εννέα ευρωπαϊκές χώρες η θυματίωση, αλλά και άλλες. Επίσης, βλέπουμε να έχουμε περιπτώσει των 100 200.000 ε, κρουσμάτων, όπως το Μαρόκο. Βλέπετε επίσης τα δεδομένα και πώς τα έχουμε καταγράψει για την περιοχή της Ευρώπης από τις εθνικές ε, έρευνες. Δυστυχώς σε κάποιες από τις χώρες έχουμε 75% ε, εξέλιξη της πρώτης μορφής φυματίωση στη δεύτερη, της MDRDP. Εάν δείτε το μέσο όρο στην Ευρώπη, την όλη δηλαδή περιοχή της Ευρώπης και τον, το παγκόσμιο ποσοστό, τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχουμε δύο σημαντικέ ε, παραμέτρου για τη θυματίωση. Το πρώτο είναι η μετανάστευση, όπου βλέπετε το ποσοστό κρουσμάτων ε, θυματίωση σε χώρε όπου καταγράφονται τα κρούσματα. Βλέπετε ότι στι περισσότερε δυτικέ χώρε, πάνω από τι μισέ ε, περιπτώσει αφορούν μετανάστε. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να σκεφτούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διασυνοριακή παρακολούθηση τη υγεία. Καθώ μετακινούνται οι πολίτε από τη μια χώρα στην άλλη, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχή υγειονομική περίθαλψη. Μια άλλη σημαντική παράμετρο είναι οι φυλακέ. Εάν δείτε τι συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, έχουμε πολλά ποσοστά θυματίωση ε, στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ένα στου δύο έχουν ενεργόμορφη θυματίωση από του ε, φυλακισμένου. Και στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε 20% περισσότερο, ε, περισσότερες περιπτώσεις ε, θυματίσεως από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ποια είναι τώρα η υπόκρισή μας ε, από τον ΠΟΗ το 2007, οι Υπουργοί Υγείας Οικονομικών, ε, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συγκεντρώθηκαν για να καταρτήσουν έναν κοινό δικό χάρτη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της DRTB. Έχουμε μάλιστα και ένα σχέδιο για την εκρίζωση της θυματίωσης και ήδη ο στόχος μας είναι να υπάρχει διαφυροποιημένη πρόσβαση στην ε, ιατρική περίθαλψη για την MDRTB, αυτή τη μορφή της θυματίωσης. Πάντως ξέρουμε ότι αυτή η μορφή είναι αυτή που θα είναι πιο διαδεδομένη στο μέλλον και γι' αυτό λαμβάνουμε από τώρα τα μέτρα μας. Τώρα την περίπτωση της Ρουμανίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τις ε, χώρες ε, της ε, περιοχής της Ευρώπης που είναι 53 και τις χώρες του ΕΟΧ. Βλέπετε ότι ο μέσος όρος στη Ρουμανία είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ ψηλότερος από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης είναι σημαντικό το ποσοστό θνησιμότητας οι ασθενεί στη Ρουμανία έχουν έξι φορέ περισσότερε πιθανότητε να πεθάνουν από θυματίωση από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το τι γίνεται με την αγωγή, η οποία είναι πολύ δαπανηρή. 500 ευρώ για τα πρώτα στάδια της αγωγής του για τον ασθενή. Εδώ βλέπετε προγράμματα που έχουν ξεκινήσει για διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ρουμανίας όπου η ομάδα ασθενών που εξετάστηκε το δείγμα είναι πολύ μικρό, 300 ασθενεί. Τα αποτελέσματα τα πρώτα είναι αρκετά ε, θερεντικά, το 70% θεραπεύτηκαν, διότι όσοι είναι εκτός ε, δεν... Ε, βλέπουμε ότι όσοι δεν ακολούθησαν την αγωγή του προγράμματος είχαν χαμηλότερα ποσοστά, να, χαμηλότερα, μικρότερες πιθανότητες να θεραπευτούν. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε εθνικά προγράμματα δράση για τι ε, χώρε τη περιοχή Ευρώπη. Στην Ρουμανία δημιουργήθηκε ένα τέτοιο εθνικό πρόγραμμα, το οποίο υποστήριξε και ο Υπουργό Υγεία και αν υλοποιηθεί, θα μπορούμε να καλύψουμε 4.500 περιπτώσεις κρούσματα MDRTB και θα εξοικονομήσουμε 250 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Θα ε, μετριαστεί ο αντίκτυπος της νόσου. Μια φωτογραφία τώρα, η οποία έχει τραβηθεί στη Ρουμανία, με τον Πρωθυπουργό τη Ρουμανία, τον ε, περιφερειακό μα διευθυντή που βλέπετε στα αριστερά, τον πρώην Επίτροπο Ντάλι, μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι η στιγμή που αποφασίζεται η υλοποίηση του προγράμματο. Να σα ευχαριστήσω και ευχαριστώ και του συναδέλφου που συνέβαλαν στη συλλογή αυτών των στοιχείων. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερω. Πρόεδρο, Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του θέματος, πολύ ενημερωτική. Και θα δώσω τώρα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιάνν Πέλα λέγομαι, δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση EuroPaid ε, διαχειριζόμαστε τις ε, συνεισφορές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Ταμείο και είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπώ την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουν και άλλα κράτη-μέλη, Πορτογαλία, Ισπανία, Φιλανδία κτλ. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Παγκόσμιο Ταμείο για να καταπολεμηθεί η φυματίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα. Πριν μιλήσω για αυτό, θα ήθελα να σας μιλήσω για το πλαίσιο για να έχουμε καλό πρόγραμμα ελέγχου της φυματίωση, ε, πρέπει να έχουμε καταρχάς ε, ένα καλό σχέδιο. Ε, πρέπει να έχουμε το τεχνικό, την τεχνική δυνατότητα Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο εκτελεί αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα και κυρίως πρέπει να δεσμευτούμε να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε ότι θα εφαρμόσουμε. Και φυσικά επαρκείς οικονομικούς πόρους, αλλά επίσης σημαντικό για τη θυματίωση, αλλά και για το AIDS, για την ελονοσία, να συνεργαζόμαστε με το πληθυσμό ή με τμήματα του πληθυσμού που είναι περιθωριοποιημένα και επομένως είναι βάλλοντα ε, και μπορεί να πάθουν αυτές τις αρρώστιες για τη φυματίωση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε με φυλακισμένους, φτωχού και με τους τσιγκάνους που γενικά είναι πολύ ευάλωτοι σε τέτοιες μολύνσεις. Επίσης, αυτοί που λένε ότι θα εκτελέσουν αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να λογοδοτούν και πολιτικά αλλά και τεχνικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχουμε διάφορους μηχανισμούς στήριξης ούτως ώστε να προωθήσουμε τον έλεγχο, καταρχάς τα εθνικά συστήματα υγείας. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ευθύνη για οργάνωση συστημάτων ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις εξωτερικές πολιτικές. Αυτός έτσι το κάνουμε, θα ρίνουμε τις χώρες να αναπτύξουν καλά ε, συστήματα υγείας με επαρκείς πόρους ε, προσπελάσιμα από όλους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι χώρες όπου έχουν υψηλά ποσοστά αφηματίωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα διαφορετικά ταμεία και σε πιο συγκεκριμένα, πιο περιορισμένα προγράμματα δημόσιας υγείας, ε, ερευνητικά προγράμματα επίσης που θα πρέπει να έχουν ε, επαρκείς πόρους για να ερευνήσουν ε, την φυματίωση για την τεχνική υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο στη Στοκχόλμη για τον έλεγχο των ασθενειών που ξεκίνησε το 2008 με ένα σχέδιο δράσης για να καταπολεμήσει τη θυματίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένο δηλαδή πρόγραμμα. Και έχει και ένα προϋπολογισμό για τεχνική βοήθεια για τις χώρες μέλης χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά εκείνε που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και υπάρχουν και διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα εθνικά συστήματα υγεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, που είναι η κύρια οργάνωση, και έχουμε και μια εταιρική σχέση ε, για θέματα φυματίωσης. Ε, υπάρχει χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της φυματίωσης ξεκίνησε μια πρωτοβουλία το 2001 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο G8 για ένα μηχανισμό χρηματοδότησης για να αντιμετωπίσουμε τις κατεπίγουσες ανάγκες κάποιων ανθρώπων φτωχών με νέα φάρμακα, κυρίως ε, ξεκίνησαμε με το AIDS που τα είχαμε στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά όχι στις φτωχότερες χώρες. Ε, ήταν σημαντικό να δοθεί αυτή η θεραπεία ε, με, σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, ε, να είναι προσιτή οικονομικά. Και αυτή η σημασία της παγκόσμιας αλληλεγγύης, αυτή η διάσταση της παγκόσμιας αλληλεγγύης δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Υπάρχουν και άλλες παγκόσμιες χρηματοδοτήσεις πέρα από το Παγκόσμιο Ταμείο. Το Παγκόσμιο Ταμείο ε, δίνει τους περισσότερους σπόρους του για το AIDS. Παρ' όλα αυτά, ε, εξασφαλίζει μόνο το 21% της διεθνούς χρηματοδότησης, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλονοσία το 5% του της χρηματοδότησης του Ταμείου εξασφαλίζεται εκεί και για την Ελλονοσία κυρίως το Παγκόσμιο Ταμείο δίνει τη χρηματοδότηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητή ε, στο Παγκόσμιο Ταμείο. Ε, συνεισφέρει πάνω από το 50% των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια, δίνει 100 εκατομμύρια το χρόνο. 110 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υπάρχουν και διάφορα μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας που χρηματοδοτούν επίσης τέτοια προγράμματα. Υπάρχει και αναπτυξιακή βοήθεια επίσης του ΟΣΕ, του ΟΣΑ, ούτως, ούτως ώστε το 0,7% του ΑΕΠ να, να δοθεί στην αναπτυξιακή συνεργασία. Οι επιμέρους δωρητές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτος και μεγαλύτερος. Εν συνεχεία βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που Ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές, Ιταλία, Ισπανία, εν συνεχεία. Συνεισέφεραν στις αρχές της δημιουργίας του Παγκόσμιου Ταμείου αρκετά έντονα, αλλά λιγότερο τις τελευταίες, το τελευταίο καιρό και έχουμε και χώρες μικρότερες σε μέγεθος, αλλά που συνεισφέρουν και αυτές Ε, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Υπάρχει κρίση χρηματοδότηση στο Παγκόσμιο Ταμείο. Ξέρετε πώς το βλέπετε. Όπως σας είπα, η αύξηση των κονδυλίων από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Ταμείο το 2001 ε, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Αυτή η μεγάλη μείωση ή μάλλον Έχουμε τήσια χρηματοδότηση. Δώσαμε σε φτωχές χώρες 3, 3, το χρόνο φτάσαμε το 2010 και το 2011 υπήρχαν προβλήματα διαχείρισης ε, στο Παγκόσμιο Ταμείο, επομένως χρειάστηκε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στο Ταμείο αυτό. Ε, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν. Το 2011 μειώθηκε κατά 2,7% η εκταμίευση, αλλά φέτος οι εκταμιεύσεις ε, θα ξαναφτάσουν πάνω από τα 3 δις και θα αυξηθούν περαιτέρω παρότι με μικρότερο ρυθμό τα επόμενα δύο χρόνια. Φτάνουμε σε ένα οριζόντιο τώρα επίπεδο, σε μια οριζόντια γραφική παράσταση. Ε, δηλαδή Κάθε χρόνο το Παγκόσμιο Ταμείο θα δίνει πάνω από 3 δις το χρόνο, αλλά δεν θα βλέπουμε αυτή η μαζική αύξηση που είδαμε τα τελευταία 10 χρόνια και είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε παρόμοιες αυξήσεις βραχυπρόθεσμα. Πάντως δεν υπάρχει κρίση με την έννοια ότι θα έχουμε μικρότερη χρηματοδότηση, λιγότερα κονδύλια από το Παγκόσμιο Ταμείο δηλαδή. Τώρα ποιος παίρνει τα πολλά λεφτά τα περισσότερα λεφτά πηγαίνουν για το AIDS. Ελονοσία, 6,5 δις και, ελονοσία, και χρηματίωση 3,8. 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι ελέγχονται 270 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει ε, θεραπεία και 3,6 εκατομμύρια παίρνουν αντιρετροϊούς για το AIDS. Η συνολική εικόνα καλή είναι. Παρ' όλα αυτά η πρόοδο είναι άνηση μεταξύ των χωρών. Σε πολλές χώρες έχουμε πρόοδο, αλλά υπάρχουν προβλήματα σε αφρικανικές χώρες. Περιορισμένη πρόοδος εκεί θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την Αφρική. Αν δούμε τώρα την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι παίρνουν κονδύλια από το Παγκόσμιο Ταμείο, με βάση το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το AIDS, αυτή τη στιγμή η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθως δεν ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο Ταμείο, αυτή είναι η πρακτική. Η Εστόνια, Εστονία ε, Πήρε 10 εκατομμύρια, αυτό ήταν μέχρι το 2007. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία ακόμα παίρνουν λεφτά από το Παγκόσμιο Ταμείο. Συνολικά έλαβαν 65 εκατομμύρια κάθε μία και αυτά τα ποσά τώρα ε, θα σταματήσουν να τα παίρνουν το 2014 και 2015. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η Βουλγαρία συνολικά έχει αυξήσει το κονδύλι της υγείας από το 9,1% στο 9,8% ε, τα τελευταία 8 χρόνια και έχει μειώσει τους εξωτερικούς πόρους που παίρνει για την υγεία από το 1,9% στο 0% ουσιαστικά. Υπάρχει μια στρατηγική ε, εφηματίωση τα επόμενα τρία χρόνια που κόστησε 37,4 εκατομμύρια. Η συνεισφορά του Παγκόσμιου Ταμείου είναι 5,2 εκατομμύρια, αλλά έχει σταματήσει εκεί. Έχει για φέτος η κυβέρνηση θα καλύψει το 60% του ετήσιου κόστους τη της δράσης για τη φυματίωση και η συνεισφορά της κυβέρνησης θα φτάσει το 15% το 100% όταν σταματήσει την χρηματοδότηση το Ταμείο. Το ίδιο ε, για το AIDS. Για τη Ρουμανία τώρα έχουμε σημαντική αύξηση σε κονδύλια από, την, από το κράτος ε, προς την υγεία από το 9,1% στο 10,8% του προϋπολογισμού οι εξωτερικοί πόροι συνεισέφεραν στο 5,7% των συνολικών δαπανών για την υγεία το 2000 και τώρα το 2009 έφτασε στο 0%. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, όπως υπόθηκε, για να διαχειριστούμε την πολυανθεκτική θυματίωση με τη βοήθεια του ΠΟΗ ε, και το Παγκόσμιο Ταμείο συνεισφέρει 3,7 εκατομμύρια. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτήν την κοινή επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Περιφερειακός Διοικητής του ΠΟΗ για την Ευρώπη ήρθε σε επαφή με τον, όχι μόνο με τον Υπουργό Υγείας, αλλά και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει αυτό το εθνικό πρόγραμμα και όταν σταματήσει να συνεισφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο, θα αναλάβει η Ρουμανία να καλύψει αυτή τη χρηματοδότηση και να Δεσμεύτηκε επίση ο Πρωθυπουργό ότι θα ενισχύσει του ελέγχου. Ο Υπουργό Υγεία συμφώνησε με τον ΠΟΗ και το ECDC να συνεχιστούν αυτές οι δεσμεύσεις και θα συνεχιστούν οι επισκέψεις τα επόμενα δύο χρόνια. Ε, συγχαίρω αυτές τις δύο χώρε για την τεράστια πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, γύρω των ερωτήσεων. Ο κύριος Τανασέσκου πρώτος. Εσείς έχετε το λόγο. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότεροι από, μας, από εσάς μάλλον γνωρίζετε την θέση μου για το θέμα αυτό. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που δίδεται σήμερα να χυθεί περισσότερο φως στο θέμα, το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε στη Ρουμανία. Πρώτα ευχαριστώ τον δόκτωρα Νταρά για τη ρεαλιστική και ακριβή παρουσίαση της καταστάσεως στη Ρουμανία. Θα προσπαθήσω νομίζω μόνο να δώσω περισσότερη έμφαση σε ορισμένα από τα όσα εξήγησε ο ίδιος και θα καταθέσω και ορισμένα ακόμα στοιχεία. Η κατάσταση στη Ρουμανία μπορεί να εξεταστεί από δύο πτυχές. Αφενός το ποσοστό επιτυχίας των θεραπείων είναι περίπου 70% όπως είπατε και μόνο 20% εκτός του πλαισίου cohort με ναι, το πλαίσιο του Παγκόσμιου Ταμείου έχουν οι ασθενείς πρόσβαση σε φάρμακα που αλλιώς δεν έχουν στη χώρα. Επίσης η παραμονή σε νοσοκομείο και η θεραπεία είναι πιο ελεγχόμενα και τα αποτελέσματα είναι βέβαια πολύ καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, στις 2 Οκτωβρίου του 12, όπως είπατε εσείς κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν, Εκρίθηκε στη Ρουμανία το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Πολυανθεκτικής Φυματίωσης για 4 χρόνια 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 5,75 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για 4 έτη. Με στόχο να φτάσουμε μέχρι το 2015 σε 75% ποσοστό αποθεραπείας. Με ένα ποσοστό που σήμερα είναι κάτω από το 20%. Ο εθνικός προϋπολογισμός για την φυματίωση ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί σε 5 εκατομμύρια για το 2013. Συνολικά θα δαπανηθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της φυματίωσης και άλλα 5 για την αντιμετώπιση της πολυανθεκτικής φυματίωσης. Άρα θα διπλασιαστεί για το 2013 ο προϋπολογισμός στα 10 εκατομμύρια. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 5 εκατομμύρια για την πολυανθεκτική φυματίωση εξαρτώνται και από την έγκριση του προϋπολογισμού το Δεκέμβριο φέτος. Εάν λοιπόν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί όπως προτείνεται, όπως έχει προταθεί, σημαίνει ότι για την αντιμετώπιση της πολυανθεκτικής φυματίωσης διαθέσιμα θα είναι μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, με το μηχανισμό, με το μεταβατικό ε, χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα αρχίσει να λειτουργεί από 1η Πρώτου του 2013, η Ρουμανία θα λάβει 3,6 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 1,8 λοιπόν τον χρόνο. Τα κονδύλια αυτά θα μπορέσουν να προσφέρουν τα φάρμακα σε 300 ασθενείς, επίσης παρεμβάσεις μεταξύ των αστέγων και ορισμένα άλλα μέτρα. Ας σημειωθεί ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Ε, υπολογίζει σε 1.500 περίπου τους Ρουμάνους ασθενείς με πολυανθεκτική φυματίωση. Επίσης, η Ρουμανία δεν διαθέτει τους πόρους για να προβεί σε διάγνωση ορισμένων ασθενών, ώστε αυτό το 1.500-1.500 ασθενείς είναι μόνο σχετικό νούμερο η Ευρωπαϊκή Οργάνωση είπε ότι η Ρουμανία πρέπει να δαπανίσει 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να αντιμετωπίσει την πολυαρθεκτική φυματίωση, ώστε συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το εθνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα για την πολυαρθεκτική φυματίωση για να εφαρμοστούν αυτά χρειάζονται περίπου 8,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και εάν δεν εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός, τότε θα χρειαστεί 13,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τώρα, ερωτήσεις για την Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει εάν προτίθεται να ζητήσει την αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Παγκοσμίου Ταμείου εάν μπορεί να μας βεβαιώσει ότι ειδικά θέματα υγείας όπως η MTRTB θα αντιμετωπιστούν και από διαφθορτικά και περιφερειακά ταμεία. Επίσης, ποια είναι τα μέτρα που προβλέπει για να βοηθήσει τη Ρουμανία να διατηρήσει τα κεκτημένα, τις κεκτημένες επιτυχίες για την αντιμετώπιση δηλαδή της φυματίωσης και της ε, πολυανθεκτικής φυματίωσης στο μέλλον και αν προτίθεται να κλιμακώσει προς τα άνω την υποστήριξη προς το Παγκόσμιο Ταμείο και επίσης ποιους άλλους διάβλους μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διοχετεύσει περαιτέρω ενίσχυση για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο κλιμάκωση της επιδημίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και έχω και μια ερώτηση για τον δόκτωρα Ταρά, αν μου επιτρέπετε. Αν προβλέπει άλλες ενδεχομένε λύσεις για να αντιμετωπιστεί το κενό χρηματοδότησης για τη Ρουμανία και από τη δική του σκοπιά ποιες είναι οι κατάλληλες λύσεις για να συγκρατηθεί ο κίνδυνος και να μην διαβεί τα σύνορα. Η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις ιατρικές σχολές παραλαμβάνεται το ίδιο στους φοιτητέ ότι καλύτερη η πρόληψη παρά η θεραπεία. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες πληροφορίες από τους δύο παρεμβαίνοντες. Πρώτον, πώς ε, έχετε οργανώσει τις προσπάθειες ε, ενημέρωσης και βαστιτοποίησης, ιδίω για το AIDS. Πώς ε, την προβλέπετε την εξτατή ενημέρωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ασθενείς αλλά τα κρούσματα που παρατηρούνται δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά πολλές φορές και με τον τρόπο ζωής του καθενός. Η σε συχνά είναι μια ασθένεια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που, που οφείλεται και σε κάποιες ε, συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως ο υποσυτισμός, η κακή διατροφή. Ποιο είναι το τμήμα του πληθυσμού λοιπόν που κινδυνεύει ιδιαίτερος, ποιοι απειλούνται από τον υποσυτισμό. Βλέπουμε πόσα κρούσματα υπάρχουν στη Ρουμανία και φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει έκρηξη της φυματίωσης στην Ευρώπη παρόλο που οι τάσεις είναι τοπικές. Υπολογίζεται πάντως να υπάρξει σημαντικός αριθμός κρουσμάτων στο μέλλον. Ακούσαμε ότι το κόστος είναι υψηλό για τα φάρμακα, για την ε, αγωγή κατά της φυματίωσης ε, και για την πρόληψη του AIDS. Υπάρχουν και ιδιαίτερα φάρμακα, συγκεκριμένα φάρμακα για την πολυανθεκτική θυματίωση. Υπάρχουν όμως ε, ειδικέ μελέτες, αξιοποιητές τα κονδύλια του Ταμείου για να γίνουν έρευνες για νέα φάρμακα, φάρμακα που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτό δεν το καλύψατε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι το Παγκόσμιο Ταμείο ασχολείται και με την ελληνοσία. Διάβασα σε αμερικανικό δημοσίευμα ότι αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες έχουν ε, βρει νέο τρόπο αντιμετώπισης του, της ελονοσίας. Οι ασθενείς έχουν μια καινούργια λύση στα χέρια τους. Η εξέβρεση λοιπόν νέων λύσεων και θεραπεία της ελονοσίας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάτι αναλόγο στην Ευρώπη. Έγιναν μελέτες στην Αμαζονία συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά ε, αξιοθαύμαστα. Υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο συσχετισμό ή να έρθουμε σε επαφή με τους επιστήμονες που κατέρθησαν αυτή τη μέθοδο για να υποφεληθούμε και εμείς. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουν κατατεθεί και υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνία σχετικά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριο Ντάρα. Για το θέμα της χρηματοδότησης. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και από την πλευρά των κυβερνήσεων. Πάντως σίγουρα υπάρχει χάσμα. Ένα χάσμα που παρουσιάζεται εδώ και πολλά χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερη χρηματοδότηση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τον καθένα θα αρκούσε να δώσει 10 δολάρια για την καταπολέμηση τη ε, θυματίωση και τη ε, πολυεθνική θυματίωση. Που θα τα εξοικονομούσαμε αν δίναμε δύο για την πρόληψη. Βεβαίω, τώρα για τι μετακινήσει πληθυσμού που είπαμε και την ε, διάδοση των κρουσμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει συνεπέστερη παρακολούθηση των ασθενών. Αυτό που κάνουμε με όλους τους αρμόδιους επιθεωρητές σε εθνικό επίπεδο και τους υπουργού ε, υγείας είναι να υπάρχει υγειονομική περίθαλψη για την ενθυματίωση διασυνοριακά εφόσον γίνεται. Ένα συνολικό πακέτο για το οποίο έχει καταρριστεί και ένα έγγραφο που, για το οποίο υπάρχει γενικώ συνένεση, απλώς απομένει να υλοποιηθεί. Πρέπει να διευκρινιστούν οι νομικές λεπτομέρειες και τα στοιχεία της χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθεί. Υπάρχουν παραδείγματα όπως στο Μεξικό για, με πολύ καλούς ελέγχους διασυνοριακούς. Στην Ευρώπη δυστυχώς δεν έχουν γίνει αρκετέ προσπάθειες. Το συζητάμε με τους αρμόδιους υπουργού υγεία για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Για την κοινωνική διάσταση και τη συλλογή δεδομένων ε, από τις χώρες η φυματίωση δυστυχώς όμως δεν πλήττει μόνο τους ε, φτωχούς εδώ. Είναι μύθο αυτό που υπόθηκε, γιατί, που είναι γνωστό για τις φυλακές. Ο καθένας μπορεί να κολλήσει φυματίωση. Το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ήδη φέρει το μικρόβιο, το μικροβακτηρίδιο της φυματίωσης. Ε, Εάν οι συνθήκε διαβίωση δεν είναι αρκετά καλές, αυτό το μικροβακτηρίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί. Βεβαίω υπάρχει συσχετισμό με τι κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε, Και βεβαίω θέλουμε να βελτιωθεί και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των ασθενών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για το νέο αυτό εμβόλιο δεν είναι ακόμα αρκετά δραστικό. Είναι κυρίως αποτελεσματικότερο στις ομάδες παιδιών. Έχουν εκπονηθεί μελέτες και γίνονται προσπάθειες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε να έχουμε ένα νέο εμβόλιο μελλοντικά όμω δεν θα γίνει αυτό μέσα σε μια τριετία, γιατί πρώτα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι παρενέργειε και πώ λειτουργεί ακριβώ ένα εμβόλιο στην πράξη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται λοιπόν με του ε, ασθενεί που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη φαρμακευτική αγωγή. Αλλά και για τα κράτη υγεία και τα συστήματα πρόνοια του θέλουμε νέα φάρμακα τα οποία να είναι και αποτελεσματικά, να λειτουργούν. Δηλαδή, οι ασθενεί που αρχίζουν να λαμβάνουν μια αγωγή να την ολοκληρώνουν κιόλα για να υπάρχει θεραπεία. Χρειάζεται βεβαίω περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη. Και βεβαίω μπορούν να συνεισφέρουν επιστημονική γνώση τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Κομισιόν. Για τη χρηματοδότηση θα σας μιλήσω. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον έλεγχο της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τόσε πολλέ ευκαιρίε χρηματοδότηση. καλύτερη... Έχουμε τι περισσότερε ευκαιρίε εδώ πέρα να ασκήσουμε έλεγχο. Η βασική ευθύνη τη οργάνωση των συστημάτων υγεία είναι οι εθνικέ κυβερνήσει, τα κράτη. Αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμε στρατηγικέ ότι χρειάζονται και βιώσιμη χρηματοδότηση, σταθερή χρηματοδότηση, καθώ και η πολιτική θέληση για να υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι, για τις ασθένειες προτεραιότητες και για να υπάρξουν παρεμβάσεις εκεί που είναι σημαντικό. Μπορούμε να δούμε και τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε τα διαρθωτικά ταμεία. Είναι μεγαλύτερη ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια από αυτά. Περιφερειακά ταμεία και διαρθωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013 είχαμε 5 δις, που είναι μόνο το 1,5% του συνολικού ποσού που διαθέτουν τα διαφορετικά ταμεία. Και οι τρεις περιοχές είναι ο επενδύσεις στον τομέα της υγείας, άμεσες επενδύσεις, ε, επενδύσεις στην, στις υποδομές, έμεσες επενδύσεις που στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας που επηρεάζουν την υγεία και επενδύσεις σε τομείς που δεν αφορούν την υγεία, αλλά που έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία, ε, που είναι κοινωνικο-οικονομικές προϋποθέσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση κάποιων ασθενειών. Έχουμε λοιπόν τα διαφορετικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να το ζητήσουν οι χώρες για να λάβουν αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες που αναφέρονται, τα δημόσια προγράμματα υγείας, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλά φυσικά η χρηματοδότηση εκεί είναι πολύ ε, μικρότερη, 50 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς μεγάλα ποσά από εκεί. Δηλαδή από τα δημόσια προγράμματα υγείας ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Φυσικά η τεχνική συνεργασία, η απόκτηση γνώσεων από τους άλλους, τεχνική βοήθεια και οικονομική υποστήριξη από την ECDC, τα δημόσια προγράμματα υγείας, ε, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υγείας όπου οι εθνικοί εμπειρογνώμονε υγεία συνεργάζονται μεταξύ του και μαθαίνουν ένας από τον άλλον. Υπό το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ένα ε, σημαντικό ποσό πηγαίνει για την θυματίωση και για ασθένειε που συνδέονται με τη φτώχεια, ε, καθώς και σε ευρωπαϊκές ερευνητικέ οργανώσεις που δουλεύουν στον τομέα αυτό αλλά πρέπει να υποβάλουν ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος οι, οι χώρες, τα ιδρύματα κτλ. Αυτά για τη γενική χρηματοδότηση, για το Παγκόσμιο Ταμείο τώρα. Η Κομισιόν θα κάνει κλιμάκωση των κονδυλίων, θα αυξήσει δηλαδή, τα κονδύλια για το... Από το Παγκόσμιο Ταμείο έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε γύρω στα 300 εκατομμύρια για το, την τριετία 11-14. Η επόμενη περίοδος ξεκινάει το 2014 και οι πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαρτηθούν από τι θα αποφασιστεί στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τα κονδύλια τα οποία θα πάνε στο Παγκόσμιο Ταμείο προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Πρόκειται για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Που Τα ποσά αυτά θα πάνε στις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κατάλογο του ΩΣΑ. Δεν υπάρχουν εκεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της ODA ε, για να επενδύσει πέρα από τις, τις αναπτυσσόμενες χώρες και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Παγκόσμιο Ταμείο υιοθέτησε ένα μοντέλο προβλέψιμο, υποστηρίζει τις χώρες στη στρατηγική τους και επενδύει στις πιο φτωχές χώρες που έχουν τις περισσότερες αρρώστιες και τη μεγαλύτερη φτώχεια. Θα υπάρξει, αυτό τι σημαίνει, θα υπάρξει μείωση στην ε, χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο ταμείο που είναι χώρες μεσαίου ή υψηλού εισοδήματος και που έχουν λιγότερες ασθένειες σε σχέση με τις φτωχότερες ε, χώρες. Αυτό σημαίνει λιγότερη, λιγότερα λεφτά για την Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες οι επενδυτικές ε, στον έλεγχο της φυματίωσης και του AIDS από τα σύνορά μας. Δεν είναι θέμα αλληλεγγύης μόνο αυτό, είναι θέμα και που μας ενδιαφέρει και άμεσα για το συμφέρον μας δηλαδή. Εμείς εισάγουμε ασθενείς από τα ανατολικά, ασθενείς ε, με AIDS και θυματίωση. Επομένως έχουμε συμφέρον να ελέγχουμε τις ασθένειες αυτές στην Ανατολική Ευρώπη. Όμως το Παγκόσμιο Ταμείο υπάρχει για να ασχολείται με χώρες που δεν μπορούν οι ίδιες να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες τους. Θα συνεχίσει χρηματοδότηση και σε πιο πλούσιε χώρε, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Πρέπει να πείσουμε τώρα τι κυβερνήσει από εκεί και πέρα να θεωρήσουν προτεραιότητά του να καταπολεμήσουν αυτέ τι ασθένειε και να του δώσουμε και οικονομική υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη όταν μπορούμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και εσωτερικά, σε εσωτερικέ πολιτικέ μα και σε εξωτερικέ μα πολιτικέ με τα χρηματοδοτικά μας μέσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα με διάλογο στο εσωτερικό μας αλλά και με τους γειτονέ μας. Πρόεδρο Γκρότε, σας ευχαριστώ. Φτάσαμε και στο τέλος τώρα του γύρου ερωτήσεων και απαντήσεων. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος και τον κύριο Ντάρα καθώς και τον κύριο Πέλερ για την παρουσία σα και τις παρεμβάσεις σας. Ε, υπάρχει βέβαια πίεση στο θέμα αυτό, αλλά βεβαίως κάθε προσπάθεια κοστίζει χρήματα, κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης. Και αυτά θα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, δηλαδή οι πολιτικές μας που είναι για την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών κινδύνων για την υγεία, χρειάζονται χρηματοδότηση. Ο αγώνας θα είναι σκληρός, αλλά χρειάζεται κάθε δυνατή υποστήριξη. Ευχαριστώ καθώς και τους συναδέλφους μου για την παρουσία τους στη συζήτηση. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι τώρα εξέταση, εξέταση της εκτελεστικής πράξης για ζωοτροφές και τρόφιμα μετά το αχυτήχημα στην Ιαπωνική Φουκουσίμα έχουμε και κροατικά ε, σήμερα και έχουμε μία ώρα και 20 λεπτά περίπου. Ας χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο αυτό που έχουμε στη, στην, ε, ε, στη διάθεσή μας. Εσείς νομίζω ε, αντικαθιστάτε την αρμοδία συνάδελφο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά, ζητώ συγγνώμη από τους Κροάτες ε, διερμηνείς. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα πλέον βασικά. Στο όνομα των Πρασίνων επιθυμώ να καταθέσω ένσταση σήμερα για την εκτελεστική πράξη που επιβάλλει ιδιαίτερες συνθήκες για τις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνικής Φουκουσίμα που είναι και στο αντικείμενο της σημερινής συζητήσεως. Τώρα η αυτή βασίζεται σε δύο σημεία και στην ουσία και στον τύπο για την ουσία δεν δεχόμαστε την πρόταση να μειωθούν οι απαιτήσει για τη δειγματοληψία και τους άλλους ελέγχους σε ορισμένα μόνο προϊόντα από ορισμένες μόνο ε, επαρχίες ή διοικητικά διαμερίσματα ιαπωνικά. Οι ε, πυρογνώμονες που μας έδωσαν ε, συμβουλές μας εξήγησαν συγκεκριμένα την κατάσταση των αντιδραστήρων της Φουκουσίμα και από το λόγο αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και ότι τελεί υπό έλεγχο. Δεν, δεν, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες εκκλήσεις ραδινεργολικούς στο περιβάλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ ε, πρόημο να ελαφρυνθούν οι περιορισμοί καθώς και οι δειγματοληπτική έλεγχοι σε προϊόντα που έρχονται από την Ιαπωνία. Από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι έλεγχοι σε όλα τα προϊόντα που ενδεχομένω είναι μολυσμένα και σε όλα τα διοικητικά διαμερίσματα ώστε να ελέγχονται ε, τα ε, πυρηνικά απόβλητα, τα ραδιενεργά απόβλητα και η ενδεχόμενη μόλυνση των ε, προϊόντων αυτών. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη σταθερότητα των αντιδραστήρων τη Φουκουσίμα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε την μείωση των ε, ελέγχων, άρθρο 10, ούτε και την τακτικότητα, τα περιοδικότητα δηλαδή της υποβολής εκθέσεων ε, στην Κομισιόν που βασίζεται στην ε, πρόταση του Φεβρουαρίου του 2012 για την ασφάλεια για τη διατροφική ασφάλεια. Το οικείο άρθρο επιβάλλει την υποχρέωση, κατά τη γνώμη μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει κάθε μέτρο για την πρόληψη κάθε κινδύνου στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν μειώνει σαφώς το επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρώσεις της, ότι η Κομισιόν υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της. Ε, η δεύτερη πτυχή της ενστάσεως που υποβάλλω στο όνομα των Ευρωπαίων Οικολόγων είναι κάπως πιο τεχνική, αλλά ελπίζω ότι θα λάβω ε, μια απάντηση πιο ορητή και ξεκάθαρη από την Επιτροπή. Η εκτελεστική πράξη υποβάλλεται στον έλεγχο του άρθρου 5 του, ε, του ε, κανονισμού 182 του 2011. Σύμφωνα με το οικείο άρθρο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να πάσα στιγμή να υποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κατά τη γνώμη του πρόταση εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες και σε τέτοια περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναθεωρήσει την εκτελεστική πράξη λαμβάνοντα υπόψη την θέση που έχει χάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οφείλει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώ και το Συμβούλιο εάν προβλέπει να διατηρήσει, τροπολογήσει ή αποσύρει την εκτελεστική πράξη. Εν προκειμένου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έσχε την ευκαιρία ούτε να αντιδράσει ούτε να υποβάλει ένσταση σε πρόταση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 11 που προανέφερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε το χρόνο να αντιδράσει στην πρώτη πρόταση διότι αυτή εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου και η μόνιμη ε, ε αντιπροσωπεία το ε, ενέκρινε λίγο αργότερα και αρχίζει να εκτελείται από το τέλος Οκτωβρίου. Εγώ βρίσκω ότι είναι λυπηρό, να μην πω απαράδεκτο, ότι δεν ε, τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Συνεπώς, μπορείτε σας παρακαλώ να μας πληροφορήσετε σχετικά με την συνέχεια που προτίθεστε να δώσετε στην σήμερα υποβαλόμενη ένσταση και εάν προβλέπετε ότι αυτή θα εξεταστεί από μέρους σας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία Ολβίε. Ε, οι τόνοι σας ανέβηκαν στο μεταξύ, μετά κατέβηκαν πάλι. Ας ακούσουμε τώρα την, άποψη, την απάντηση μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ... Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Και εγώ θα βάλω τους κουράδες εκεί διερμηνείς να δουλέψουν. Nous étions dans une euh, η νομική μας κατάσταση ποια ήταν. Ο προηγούμενος κανονισμός της 29ης Μαρτίου 2012 εξέπνε την 1η Νοεμβρίου του 2012. Δηλαδή, αν δεν γινόταν τίποτα, αν η Κομισιόν δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία πριν την 1η Νοεμβρίου του 2012, τα παλιά μέτρα ξαφανίζονταν και επομένως δεν θα υπήρχε κανένα μέτρο ελέγχου και στην αφετηρία και στην άφηξη των Ιαπωνέζικων προϊόντων. Μπορούσαν να μπουν δηλαδή ωραιότατα, χωρίς κανέναν έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν δεν θελήσαμε να, μπούμε, να δεχτούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή να ζήσουμε μια κατάσταση όπου θα μπαίναν τα προϊόντα χωρίς ελέγχους. Συζητήσαμε με τις Ιαπωνέζικες Αρχές το θέμα, που θέλανε πιο ελαστικούς ελέγχους φυσικά, αλλά περιμέναμε και τα τελευταία αποτελέσματα από την τελευταία σοδιά οποροκυπευτικών και ρυζιού, ας πούμε. Το καλοκαίρι ήταν αυτή η τελευταία σοδιά. Γι' αυτό λοιπόν παρουσιάσαμε αυτό το σχέδιο απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το στείλαμε στις 10 Οκτωβρίου ψηφίστηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή και υιοθετήθηκε σύντομα στις 26 Οκτωβρίου με την ε, ταχεία διαδικασία πριν την διαβόητη 1η Νοεμβρίου. Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης του παλιού κανονισμού, της παλιάς νομοθεσίας τέλος πάντων, θελήσαμε να υιοθετήσουμε ένα μέτρο σύνεσης και αναλογικό. Να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από τη μία του καταναλωτή, από τις εισαγωγές ιαπωνέζικών προϊόντων. Φυσικά η κατάσταση των αντιδραστήρων της Φουκουσίμα, ανάλογα με το ποιος θα εξετάζει, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υποέλεγχο και ή δεν είναι υποέλεγχο. Δεν ξέρουμε αν θα βελτιωθεί ή θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Οι Ιαπωνέζικες αρχές μας λένε ότι η κατάσταση είναι υποέλεγχο και μας απέδειξαν με πολλές δοκιμές, με πολλά πειράματα, ότι, παίρναν, ότι τα έβλεπαν τα πράγματα πολύ σοβαρά. Μετά το ατύχημα του Μαρτίου του 2011, οι Ιαπωνέζοι έκαναν πάνω από 300.000 τεστ σε διάφορα τρόφιμα που παράγονται στα διάφορα διαμέρισματα της χώρας και κυρίως στη Φουκουσίμα. Από τις αρχές του 12 τώρα έκαναν 167.000 τεστ. Διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου για όλα αυτά τα τρόφιμα. Κυρίως για την εγχώρια κατανάλωση, προφανώς, αλλά και για τις εξαγωγές. Γιατί ξέρετε ότι πρέπει να κάνουν ελέγχους πριν τις εξαγωγές από τις 12 περίφημες περιοχές τους. Τώρα, τα κράτη-μέλη από τις 11 Μαρτίου και μετά έκαναν περίπου 3 εκατομμύρια τεστ. Πέρα από τις ε, δοκιμές και τεστ που κάναν οι Ιαπωνέζοι πριν την εξαγωγή. Τον Ιούνιο του 2011, πάνω από ένα χρόνο που η Γαλλία ανακάλυψε δύο παρτίδες τσαγιού μολυσμένου, δεν έκανα τίποτα. Σε όλα προϊόντα είχαμε θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, λογικός πώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στους, στους Ιαπωνέζους και στα τεστ που κάνουν εκείνοι. Με αυτό το νέο μέτρο τώρα προβλέπονται κάποιες αλλαγές σε σχέση με την παλιά κατάσταση για δύο διαμερίσματα όπου μειώσαμε τους ελέγχους, αλλά τους διατηρούμε για ένα στα μανιτάρια και το τσάι και για το άλλο μόνο για, το... για τα μανιτάρια. Γιατί ξέρετε ότι στα μανιτάρια συγκεντρώνται τα ενεργά στοιχεία. Τώρα για το διαμέσμα της Φουκουσίμα. Κρατήσαμε τα μέτρα που υπήρχαν ήδη. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε όλα τα τρόφιμα, εκτός από το τα ενοπνευματόδη. Αλλά για όλα τα τρόφιμα υπάρχει έλεγχος. Και για τις εννέα άλλες περιοχές, από τις 12, Υιοθετήσαμε ένα κατάλογο 41 προϊόντων σε σχέση με τον παλιό κατάλογο που ελέγχαμε όλα τα τρόφιμα. Ο κατάλογος αυτών των 41 προϊόντων που πρέπει να ελέγχουν οι Ιαπωνέζικες αρχές πριν από την αποστολή των τροφίμων, εκεί εντάσσονται τα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ε, περιλαμβάνονται εκεί προϊόντα βραχίας ζωής, όπως σαλάτες και λαχανικά που τα κρατάμε δύο, τρεις, τέσσερις μήνες. Που ξέρουμε ότι τα καλλιεργήσαμε σε περιοχές καθαρές, χωρίς ραδιενέργεια. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είναι ραδιενεργά γιατί δεν, ε, δεν τους επικάθησε ραδιενεργή σκόνη το Μάρτιο του 2011. Και μια και η περίοδος καλλιέργειας είναι σύντομη, θεωρήσαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να μπουν σε αυτόν τον κατάλογο. Κρατήσαμε όμω τα 41 αυτά προϊόντα στον κατάλογο. Επίσης, έχουμε μια συχνότητα ελέγχου ύψου 5% για όλα τα διαμερίσματα αυτά. Όχι τα 12 μόνο, για όλα. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχων πέρα από τους πολλαπλούς ελέγχους που κάνουν οι Ιαπωνέζοι. Υπενθυμίζω ότι πέρα από τις δύο αυτές παρτίδες της Αγίου του Ιουνίου 2011, μετά τον Ιούνιο δεν είχαμε ποτέ κρούσματα, ποτέ πρόβλημα ραδιενέργειας σε τρόφιμα. Συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε. Τα μέτρα που υιοθετήσαμε είναι αναλογικά, είναι προσαρμοσμένα στην κατάσταση και στη βελτίωση της κατάστασης ήδη στην Ιαπωνία. Δεν αλλάξαμε τους κανόνες. Έχουμε κρατήσει τους γιαπωνέζικους κανόνες που είναι πολύ πιο αυστηροί από τους ευρωπαϊκούς. Κανόνες που εμείς έχουμε από το Τσερνομπίλ. Οι Ιαπωνέζοι έχουν για τον εαυτό τους αυτούς τους κανόνες πιο αυστηρούς και τους έχουμε κρατήσει. Και μάλιστα τους είχαμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες. Επιβάλαμε αυτούς τους ε, Ιαπωνέζικους κανόνες που είναι οι πιο αυστηροί στον πλανήτη. Επίσης δεν έχουμε υπερβεί τις αρμοδιότητές μας, απαντώ στην ερώτησή σας εδώ. Στα πλαίσια του άρθρου 53 του General Food Law έχουμε κρατήσει τα πιο σημαντικά μέτρα, τα έχουμε προσαρμόσει στη σημερινή κατάσταση σε σχέση με το ατύχημα που έγινε πριν από 1,5 χρόνο. Είναι σαφές τώρα ότι αν οι αντιδραστήρες λιώσουν, αν αρχίσουν να εκλείουν ραδιενέργεια και να μολύνουν το περιβάλλον, φυσικά θα πάρουμε τα, κατα... τα αντίστοιχα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό. Ζούμε στο παρόν. Μέσα σε 24 ώρες μπορούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία και να την προσαρμόσουμε σε νέα δεδομένα. Αν υπάρξει ραδιενεργή μόλυνση λόγω οποιοδήποτε προβλήματος στους αντιδραστήρες. Θεωρούμε λοιπόν ότι προσαρμοστήκαμε στην κατάσταση. Αλλιώς το μέτρο θα εξέπνε την 1η Νοεμβρίου. Και δεν θα είχαμε τίποτα στη διάθεσή μας. Δεν θεωρούμε ότι ξεπεράσαμε τις αρμοδιότητές μας. Χρησιμοποίησαμε τα δεδομένα και προσαρμοστήκαμε στην κατάσταση. Αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν. Φτάσαμε στο τέλος της ημερησίας διατάξεως και τι να πω. Εύχομαι στις συναδέλφους καλό βράδυ καθώς και στους εκπροσώπους της Κομισιόν. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 17 και 18 Δεκεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες και θα προσκαλέσω όλες τις συναδέλφους, βέβαια και οι άρενοι συνάδελφοι μπορούν να προσέλθουν αν θέλουν, στις 17 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, στις 8 το βράδυ, σε μια μικρή δεξίωση της επιτροπή περιβάλλοντο με την ευκαιρία των Χριστουγέννων θα υπάρχει κάτι, ε, θα υπάρχουν και κάτι ε, που θα μπορεί κανείς ε, να πιει και τα σχετικά και εδώ κλείνω τη συνεδρίαση και σας εύχομαι καλή επάνωδο ή πάντως καλή ανάπαση.